Um, λοιπόν, συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω στην εξαιρετική αυτή συνεδρίαση για το δίκαιο του καναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεταφορά και την εφαρμογή του στο, εθνικό, στο εθνικό δίκαιο και είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για κοινή συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια. Αναμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και τη δική σας εμπειρία και διαλέξαμε να εξετάσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς νομίζουμε ένα από τα σημαντικότερα, μια από τις σημαντικότερες αλλαγές ε, στην θητεία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πλησιάζει στο τέλος της και λάβαμε την πρόταση οπότε θέλω να το συζητήσουμε να ακούσω τις απόψεις σας ε, και να μπούμε μετά στις λεπτομέρειες. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σας παρακαλώ να εκφραστείτε ελεύθερα. Και βεβαίω καλωσορίζουμε και τον κύριο Γίλεκ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Μεταφορών ε, της Γερουσίας της Τσεχίας ε, και βεβαίως ε, και εκείνος θα σας καλωσορίσει γιατί αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την Τσεχική Προεδρία για πολλούς φακέλους που περνάνε από την Επιτροπή μας. Έχετε λοιπόν τον λόγο, κύριε Γιλέκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της ε, γερουσίας ε, της Τσεχίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ σήμερα γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερα το δίκαιο των καταναλωτών. Το δίκαιο των καταναλωτών στην Τσεχία και σε πολλά άλλα από τα νέα είναι μια καινούργια υπόθεση, ακόμα αναπτύσσεται, δεν είναι κάτι τόσο παλιό σωστά παλιά κράτη-μέλη, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας εξουλούν αυτά τα ζητήματα, γιατί η προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα και των ευδηματιών ε, είναι πολύ σημαντικά, ειδικά όταν μιλάμε για απέμπτες εμπορικές πρακτικές. Και βεβαίως όλα αυτά μας βοηθούν πάρα πολύ. Είναι λοιπόν σημαντικό να επικεντρωθούμε στο σωστό εμπόριο και να έχει και υψηλής ε, ποιότητας υπηρεσίες ο καταναλωτής. Επίσης ε, χαίρομαι για την ε, παρουσία σας στην αίθουσα και ελπίζω να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ε, ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος της συνεδρίασής μας. Να σας υπενθυμίσω τον κανονισμό του Κοινοβουλίου που ίσως διαφέρει από τα δικά σας κοινοβούλια. Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα έντυπο για να ζητήσετε το λόγο, θα τα δώσετε μετά στους κλητήρες και θα τα δώσουν σε μένα. Νομίζω το καλύτερο είναι αυτό γιατί δεν βλέπω τα ονόματά σας ε, μπροστά μου, οπότε συμπληρώστε το όνομά σας ε, για να σας δώσω τον λόγο για την παρέμβασή σας. Όπως είπα, περνάμε στο πρώτο μέρος. Αυτό το οποίο ήθελα να κάνω είναι να σας υπενθυμίσω πως η κυρία Κούνεβα θα έρθει σε λίγο. Ήθελα να ξεκινήσουμε για να προχωρήσουμε εμεί, Οπωσδήποτε θα καλωσορίσουμε την κυρία Κούνεβα όταν έρθει. Το πρώτο μέρος λοιπόν της συνεδριασής μας είναι η τρέχουσα συζήτηση και ξέρω ότι πολλοί θα τα συζητάτε αυτά και στα δικά σα κοινοβούλια. Η οδηγία δικαιωμάτων του καταναλωτή και οι μελλοντικέ εξελίξεις στο δίκαιο των καταναλωτών. Εμεί στην Επιτροπή αυτή οπωσδήποτε θεωρούμε πως είναι εξαιρετική στιγμή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 η διερμηνία. Μα συγχωρείτε για το, τεχνικό πρόβλημα. Επανήλθε η διερμηνία πάντως. Μα συγχωρείτε, προς στιγμή αναβόζησαν τα μηχανήματα. Yes, okay, Ήρθε και η κυρία Επίτροπος. Έχετε διερμηνία, ακούγεται η ελληνική διερμηνία, παρακαλώ. Ωραία. ξεκινήσουμε ξανά. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κούνεβα που δραστηριοποιείται πολύ στην ε, προστασία των καταναλωτών. Η Επιτροπή μας εργάζεται εντατικά και έχουμε συχνές συναντήσει με την κυρία Κούνεβα, οπότε χαίρομαι που ήρθε και σήμερα. Ας ξεκινήσουμε ελπίζω με διερμηνία αυτή τη φορά. Όπως σας είπα, καλούμεθα να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα και για τους καταναλωτές στη σημερινή οικονομική κρίση. Θέλουμε απλούστερους κανόνες για τις επιχειρήσεις για να μπορούν να προσφέρουν προϊόντα αγαθά και υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά χωρίς να μειώνεται η προστασία των καταναλωτών και χωρίς ε, προστασία των καναλτών δεν θεωρούμε ότι οι καναλτές θα μπορούν να διαλέγουν ή να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε άλλα κράτη ε, μέλη θα καταναλώνουν στην δική τους χώρα εάν ε, θεωρούν ότι δεν έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε αυτή τη στιγμή με αυτή την νομοθεσία για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά με το να βελτιώσουμε και να απλοποιήσουμε την ομοθεσία και την εφαρμογή της, κάτι που θα μας απασχολεί στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίασης. Και η πρόταση αυτή είναι μια εκβάθρον μεταρρύθμιση του δικαίου περί καταναλωτών. Γι' αυτό και στην δική μας Επιτροπή και στα Εθνικά Κοινοβούλια εξετάζουμε αυτή την νομοθεσία για να καταλήξουμε σε ένα σωστό νομοθέτημα. Όπως ξέρετε, αντικαθιστά τέσσερις υπάρχουσες οριζόντιες οδηγίες με μία ενιαία οδηγία που μας οδηγεί σε πλήρη εναρμόνιση. Και πρέπει να συμμεθυμίσω ότι με την ελάχιστη εναρμόνιση τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν τους ε, κανόνες ή να υιοθετήσουν ισχυρότερους, αλλά τώρα πλέον δεν θα υπάρχει απόκληση με την πλήρη εναρμόνιση. Και αναφέρθηκε πως ε, πράγματι οι γενικοί ε, κανόνες συμβάσεων μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν στα κράτη-μέλη. Οπότε βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη δική σας δουλειά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προσέγγιση τώρα που είχαμε 10 Νοεμβρίου αποφασίσαμε εγώ να προχωρήσω αυτή την ε, πρόταση ως πρόεδρος της Επιτροπής με τους, σύμπρο, με τους αντιπροέδρους της Επιτροπής και με τους πολιτικούς συντονιστές που μπορεί να είναι αυτό το οποίο λέμε επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας στα εθνικά κοινοβούλια. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν ο πιο συνενετικός ε, τρόπος για να προχωρήσουμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία. Επίσης αποφασίσαμε ότι λόγω της πολυπλοκότητας και του εύρους αυτής της πρότασης και του περιορισμένου χρόνου, γιατί αυτό το κοινοβούλιο τώρα θα διακόψει σε ένα μήνα για να ακολουθήσουν οι ευρωεκλογέ. δεν θέλαμε παρόλα αυτά να βιαστούμε, οπότε αποφασίσαμε να συντάξουμε αυτό το έγγραφο εργασίας με την ησυχία μας, το οποίο αποφασίσαμε θα αποσταλεί στα εθνικά κοινοβούλια, στι επιτροπές σας, για να μπορείτε να δείτε και εσείς το τι κάναμε και βέβαια θα γίνει και αναλυτική συζήτηση με την κυρία Κούνεβα στην τελευταία ολομέλεια του Μαΐου, όπου θα κατατεθεί μια προφορική ερώτηση και οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν ότι θα ήθελαν ένα ψήφισμα για το έγγραφο αυτό εργασίας και για να μας δώσουν μια ιδέα του τι θα θέλαμε να γίνει σε αυτό το φάκελο. Αυτά εν ολίγης ε, και μπορούμε να πούμε ότι προδιαγράφουμε τροχιά που θα ακολουθεί στο νέο κοινοβούλιο. Ένα από τα πρώτα ζητήματα λοιπόν που μας απασχόλησε, αφού μας το ζήτησαν αυτό η των πολιτικών ομάδων, είναι να δούμε την αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν, να ερευνήσουμε το πώς ε, Καταλήξαμε στην πρόταση αυτή που έχουμε επιτάπητο. επίση να γίνει μια δημόσια ακρόταση με όλου του ενδιαφερόμενους. Ήδη έχει γίνει μια δημόσια ανταλλαγή απόψεων, αλλά όπω είμαι σίγουρη ότι ξέρετε, το ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση είναι τόσο μεγάλο ώστε δεν μπορέσαμε να προσκαλέσουμε όλου του ε, ενδιαφερομένους. Οπότε αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική με τα νέα μέσα, να γίνει δηλαδή μια διαβούλευση μέσω διαδικτύου και να γίνει έτσι τελικά η διαβούλευση αυτή και μπορείτε και αυτό να το δείτε, μάλιστα είναι διαθέσιμο. Ήταν μια άτυπη και πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, γιατί δεν τους είπαμε μόνο τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει, είπαμε εάν δεν σας αρέσει τι προτείνετε εσείς για να προχωρήσει αυτό το, το ζήτημα, γιατί θεωρούν πως οι στόχοι της Κομισιόν είναι σωστοί, και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη σε επιχειρήσεις αλλά να έχουμε και υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Απευθυνθήκαμε και στις 27 αντιπροσωπείες των ε, κρατών μελών, τις μόνιμες αντιπροσωπείες δηλαδή που βρίσκονται εδώ γύρω στις ε, Βρυξέλλες και ζητήσαμε να απαντήσουν ειδικά στο εξής ερώτημα. Εάν υιοθετήσουν αυτή την πρόταση στο κράτος μέλος σας, τι σημαίνει αυτό για το εθνικό σας ε, δίκαιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα για τα κράτη-μέλη να βρουν δηλαδή ποια είναι τα ζητήματα τα κράτη-μέλη και να μας απαντήσουν. Γραπτός. Όπως σας είπα, θα παρουσιάσουμε το έγγραφο εργασία, θα σας το αποστείλουμε, αλλά έχει ξεκάθαρο πεδίο εφαρμογής. Ε, βλέπουμε δηλαδή την αξιολόγηση αντικτύπων, τις βασικές πτυχές της εναρμόνισης, το επίπεδο της εναρμόνισης. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για να πούν και οι συνάδελφοι κάτι, αλλά θα έχετε βεβαίως διαθέσιμο αυτό το έγγραφο εργασίας και όπως σας είπα θέλουμε να βασιστούμε και στη δική σα συνεισφορά για να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση αποτελεσματική για να έχουμε μια νομοθεσία η οποία θα προσφέρει πραγματικά στους πολίτες μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω και πάλι από τον κύριο Γιλεκνά μας πει τα της Επιτροπής. Α, πρώτα απ' όλα έχουμε, θα ακούσουμε την Επίτροπο την κυρία Κούνεβα, με συγχωρείτε. Και μετά θα δώσω τον λόγο σε εσά για να έχετε όλη την ευκαιρία να εκφραστείτε. Ε, ευχαριστώ. Thank you very much, and... Ευχαριστώ πολύ. Αιλίν, καλημέρα σε όλους. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς να συζητήσουμε δηλαδή ανοιχτά την πιο σημαντική εξέλιξη στο δίκαιο καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, καλωσορίζω ε, τη δική σας συνεισφορά και ελπίζω να μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να μην Λυσμονούμε όμως ότι υπάρχει ήδη κείμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει. Και θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή στα κράτη-μέλη, ε, που από ό,τι έχω καταλάβει ε, αφιερώνεται τη δεύτερη συνεδρίαση σήμερα. Και πώς είναι ε, δυνατόν να δικαιώνονται οι καταναλωτές κάθε φορά. Από τότε που ανέλαβα φρόντισα να υπάρχουν υγιείς ε, αγορές, καλώς λειτουργούσες, να έχουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη οι ε, καταναλωτές και όταν έχουμε διασυνοριακά ε, συνεργασία και εμπόριο και καινοτομία αυτά να ενθαρρύνονται. Αγωνιστικές αγορές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία Υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει για την ενιαία αγορά για να λειτουργεί καλύτερα για όλους μας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο τα δικαιώματα των καταναλωτών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ακριβώς επειδή είναι κατακαιρματισμένα όλα αυτά και ε, υπάρχει και η Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης, ένα δεν γνωρίζετε, κάθε κράτος μέλος, ε, αν θέλει κάποιος μάλλον να πουλήσει κάποια προϊόντα σε μια άλλη χώρα θα πρέπει να συμμορφωθεί και να προσαρμοστεί σε 27 διαφορετικές νομοθεσίες. Αυτό είναι τεράστιο βάρος για ε, τις επιχειρήσεις, όπως έδειξε και η μελέτη αντικτύπου που κάναμε. Η κρίση σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρή και επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα του νομικού κατακαιρματισμού στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Γαλλία ε, έχει κανείς δικαίωμα μία εβδομάδα να αλλάξει γνώμη, ε, μία ημερολογιακή εβδομάδα, εάν αγοράσει κάτι και δεν του αρέσει. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι 7 εργάσιμες ημέρες, ενώ στη Δανία και στη Μάλτα είναι 14 και 15 ημερολογιακές ημέρες. Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει πώ μετράμε τη μέρα, εργάσιμη μέρα ή μέρα ημερολογιακή. Και φανταστείτε τι ε, μηνύματα στέλνουμε στις επιχειρήσεις και τι προστασία και τι ασφάλεια στους καταναλωτές για να τους ενθαρρύνουμε ότι θα πρέπει να έχουν και διασυνοριακή ε, ενιαία αγορά. Γι' αυτό δεν μα εκπλήξει που καμιά φορά η έμπορη σου λέει δεν πουλάω online. Ένα στους πέντε λιανοπολιτές, 21% πουλάει διασυνοριακά σήμερα στην Ένωση. Η μισή ε, από τους υπολείπους που δεν πουλούν ε, δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να το πράξουν. Εάν το κόστος συμμόρφωσης θα περιοριστεί σημαντικά. Χτες συγκεκριμένα το απόγευμα και σήμερα το πρωί έχουμε σύνοδο κορυφής ε, των καταναλωτών για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες Έχουμε ε, ενώσεις καταναλωτών, έχουμε και επιχειρήσεις, εταιρείε και εμπόρους. Και ακριβώς αυτή η άρνηση των εμπόρων να πουλούν σε άλλη χώρα, ήδη έχει πολιτικοποιηθεί ο ζήτημα. Ιδιαίτερα πολίτες της ε, Ανατολική Ευρώπη Ευρώπης λένε, εμεί εμείς είμαστε από νέα κράτη-μέλη, μα τιμωρείτε, δηλαδή επειδή φτάσαμε αργότερα και δεν θέλετε να μα πουλάτε. Υπάρχει δηλαδή Ευρώπη, Ευρωπαίος καταναλωτής δεύτερης κατηγορίας. Όχι, εμεί ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι απλή αγορά. Και κάθε ξεχωριστό μήνυμα της αγοράς θα μπορούσε, μπορεί πάντα να ερμηνεύεται με πολιτικό τρόπο. Καταλαβαίνω ότι και οι καταναλωτές και οι έμποροι μπερδεύονται και δεν θέλουν, ε, διστάζουν να ε, εκμεταλλευτούν πλήρω το δυναμικό τη νέα αγορά. Εγώ θέλω να δράσω εκεί, αλλά θα πρέπει δύο ζητήματα πρώτα να εξετάσουμε σημαντικά. πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τη ε, λειτουργία της αγορά για τους καταναλωτέ και πώς μπορούν να υποφελούνται καλύτερα οι καταναλωτέ. Είναι να ξεκλειδωθεί η αγορά, να ανοίξει και να τονωθεί, να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ακριβώς αυτό ε, αποσκοπεί και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αποτέλεσμα ευρύτατης δημόσιας διαβούλευσης. Δεν έχει γραφτεί σε τίποτα γραφεία επιτρόπων και της Επιτροπής. Ενισχύει την προστασία των καταναλωτών με ενιαία δικαιώματα, με ίση προστασία όπου και αν αγοράζουν και με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι στο διαδίκτυο είτε στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για τους πολίτες και κάποιος που ζει στην Πράγα, στο Βερολίνο, ε, θα μπορούσε να υποφεληθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό να αγοράζει ε, από το διαδίκτυο, από την Κοπεχάγη, το Λονδίνο, ακόμα και από μια μικρή πόλη της Ελλάδας, χωρίς να ταξιδεύει. Είναι δικαίωμα του καταναλωτού η πρόσβαση στην αγορά. 30 χρόνια μας απασχολεί αυτό και πλέον έχουμε 500, 500 ε, εκατομμύρια καταναλωτές. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες πιέζονται πολύ και η εμποροί είναι δύσκολοι καιροί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Στόχος ε, είναι η αύξηση ε, της ευημερία ε, των καταναλωτών. Βεβαίως πάντα η οδηγία από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Μακάρι να γινότανε. Ούτε αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι πολίτες. Αλλά υπάρχουν ε, ε, ωφέλη. Για παράδειγμα, έχουμε αυστηρούς νέους κανόνες για την παράδοση. Γνωρίζουμε, γιατί το έχουμε μελετήσει, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους καταναλωτές στη διασυνοριακή συναλλαγή είναι ακριβώς αυτό. Και εντός ενός μηνός θα πρέπει να παραδίδονται τα αγαθά παντού στην Ευρώπη. Και υπάρχουν και νέοι κανόνες σχετικά με τη ζημία ή την απώλεια κατά τη μεταφορά. Γιατί σήμερα είναι σκέτη κουρελού αυτό το ε, τοπίο. Ανθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο σε κάποια κράτη-μέλη, ε, υπάρχει το πρόβλημα αυτό ε, της μη παράδοσης, μη έγκαιρη παράδοσης ή παράδοση ε, προϊόντων. Και να μην υπάρχουν ε, συγκαλυμμένα ε, δαπάνες και, και έξοδα. Δηλαδή να πληρώνει κανείς μόνο ό,τι αναγράφεται και ό,τι γνωρίζει. Επίσης να υπάρχει περίοδος περισυλλογής και αλλαγής γνώμης ε, δύο εβδομάδων και να μην υπάρχουν ε, στην online αγορά ε, κάποια κουτάκια που ήδη να έχουν εγκριθεί ως επιπλέον δαπάνες, ασφάλειες κτλ. χωρίς να το έχει κάνει ο καταναλωτής. Ανοίγει σελίδα και είναι ήδη καλυμμένα αυτά. Επίσης, δεν θα πρέπει να γίνεται άγρα πελατών. Καλύπτεται δηλαδή και όταν σου χτυπάει πλασιά την πόρτα. Ε, αυτή η περίπτωση. Κλείσαμε τα παραθυράκια για τις ε, πωλήσει εξ αποστάσεως. Όλα αυτά τα συμβόλαια καλύπτονται. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένη προστασία του καταναλωτή για χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες, ε, Βασίλειο συγγνώμη, και η Δανία. Υπάρχουν ενισχυμένε επίσης υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια θα πρέπει πάντα ο καταναλωτής να γνωρίζει όταν ε, υπάρχει κάποια εγγύηση ή ένα ποσό που δεσμεύεται στην πιστοτική του κάρτα. Να μπορεί με απλό email ε, να καταγγείλει τη σύμβαση ή η διόχειρη επιστολή ο καταναλωτής με τα δικά του λόγια. Δεν χρειάζεται εμπορική ορολογία. Υπάρχει τώρα ε, μια φαιά λίστα και μαύρη λίστα με φιλικό τρόπο προς τον πολίτη, προς τον καταναλωτή και όχι ψηλά γράμματα στα συμβόλαια. Είναι απλά λοιπόν αυτά τα πράγματα ε, για να γνωρίζει ο κλάδος και οι έμποροι. Η πρόταση αυτή ε, ε, βέβαια είναι υπέρ του καταναλωτού ή υπέρ του εμπόρου. Εγώ πιστεύω, γιατί ε, ορισμένοι λένε ότι έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και αντιασελόμενα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι είναι καλό για τον καταναλωτή, είναι καλό για τον έμπορο και ε, το αντίστροφο. Εσωτερική αγορά είναι και τους καταναλωτές θέλουμε να βοηθήσουμε. Όταν λειτουργεί μια αγορά καλά, αυτό είναι ο καλύτερος φίλος του καταναλωτού. Θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι, συνειδητοποιημένοι και να παίζουν και αυτοί ενεργά το ρόλο τους η πρόταση δεν αναγκάζει τα κράτη-μέλη να ε, καταργούν το δίκαιό τους περί συμβάσεων, το ενοχικό δίκαιο, ούτε τις εγγύσεις για τις υπηρεσίες, όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες ε, ε, των οικοδομών. Ή χρειάζεται να έχουν επιπλέον εμπορική εγγύηση. Χρειάζεται ε, ακριβώς προστασία του καταναλωτού και προστασία των εμπόρων ταυτόχρονα. Ε, έτσι υπάρχουν ευκαιρίες παντού στην Ευρώπη, ευκαιρίες και δυνατότητες προσαρμογής παλαιών συστημάτων απαρχιωμένων και αυτό τελικά έχει καλές επιπτώσεις και στις τιμές ε, και οι εταιρείε έχουν ασφαλές περιβάλλον μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να γνωρίζουν το κόστος. Ε, προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας επικοδομητική σε εθνικό επίπεδο, στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε ένα άλλο θέμα, εξίσου σημαντικό, ε, που είναι η εφαρμογή και επιβολή ε, των κανόνων προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αν δεν εφαρμόζεται σωστά και αν δεν επιβάλλεται σωστά σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στενά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε ορθά και εγκαίρω να μεταφέρονται οι οδηγίες ε, στην εθνική νομοθεσία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει η εθνική νομοθεσία, βοηθάει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τα κράτη-μέλη για να εφαρμόζουν ομοιόμορφα την νομοθεσία αυτή. Να σα δώσω σύντομα ε, κάποια παραδείγματα για τις πρόσφατες οδηγίες, μια οδηγία για θέμητες εμπορικές πρακτικές και ε, για την καταναλωτική πίστη. Τώρα για την πρώτη οδηγία έχουμε εθνική νομοθεσία σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, μόνο σε δύο δεν ε, Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να βεβαιωθούμε ότι αυτή η οι είναι σύμφωνοι με την οδηγία και όπου χρειάζεται προσφεύγουμε στο δικαστήριο και φροντίζουμε να βλέπουμε, να εφαρμόζεται και όλο η νομοθεσία και όχι απλώς να εγκρίνεται. Η ενιαία εφαρμογή σημαίνει ότι με τον ίδιο τρόπο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις ίδιες έννοιες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει αυτή η οδηγία για θέμητες εμπορικές πρακτικές να καλύπτει νέους κλάδους που εμφανίζονται τώρα στην αγορά για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για να απαντήσουμε ε, σε διαφορετικές ενδεχομένω ερμηνείες ε, στον πρώτο χρόνο προσαρμογής, στον πρώτο χρόνο εφαρμογής για να βελτιώσουμε ε, την αντίληψη και την κατανόηση βασικών όρων και νιών. Για να σας δώσω ένα σύντομο και πρόσφατο παράδειγμα της οδηγίας αυτής που εγκρίθηκε πέρσι τον Απρίλιο. Τα κράτη-μέλη ε, καλούνται μέχρι τον Ιούνιο του επομένου έτους να τη μεταφέρουν και η Κομισιόν τους υποστηρίζει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Ε, οργανώνει, μάλιστα ήδη έχει οργανώσει δύο εργαστήρια με τα κράτη-μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας, ε, το ένα τον Νοέμβριο και το άλλο τον περασμένο μήνα. Στόχος ήταν να δούμε ποια είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα, μια ιστοσελίδα σύρκα για να βελτιώσουμε τις συζητήσεις και τις ε, ε, βέλτιστες πρακτικές που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών. Για την επιβολή θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι κανόνες είναι σαφείς και ε, ισχυροί και εφαρμόζονται με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό. Οι περισσότεροι έμποροι είναι ειλικρινείς και τίμοι, αλλά ορισμένοι άλλοι που είναι κερδοσκόποι ε, έχουν και αθέμητες πρακτικές καμιά φορά και σχροκέρδια. Ε, αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμόζονται ε, σωστά. Αυτό είναι κυρίως έργο των κρατών μελών. οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να έχουν το δυναμικό που τους χρειάζεται και τις εξουσίες για να σταματούν και να τερματίζουν αυτές τις πρακτικές. Υπάρχουν και οι τεχνολογικές και οι οικονομικές δυνατότητες σήμερα πλέον με νέες ε, ευκαιρίες για να ε, δρουν σε ένα περιβάλλον διασυνοριακό όπως είναι η εσωτερική αγορά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε όλα αυτά να μεταφέρονται και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέγω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, και την καλύτερη νομοθεσία του κόσμου να έχουμε, αν δεν την εφαρμόζουμε αποτελεσματικά δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έχουν γίνει πολλά ακόμα, έχουν γίνει πολλά συγγνώμη, αλλά ε, είμαι πεπισμένη ότι πολλά απομένουν να γίνουν σε συγκεκριμένους τομείς και θα πρέπει αυτό να γίνει συντονισμένο. Στις αερομεταφορές το 2007 κάναμε έναν έλεγχο και καταλήξαμε σε ένα κατάλογο 30 σημείων σε συνεργασία με τον κλάδο και ε, είναι υποχρεωμένε οι ιστοσελίδε που πολλούν αεροπορικά εισιτήρια να συμμορφωθούν. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του έτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μελέτη για να δει σε ποιο βαθμό βελτιώθηκε η κατάσταση. Επιπλέον, ένας έλεγχος ε, υπηρεσίε κινητή τηλεφωνία έγινε επίση. έδειξε ότι 80% των ιστοσελίδων που πολλούν ringtones ή αντίστοιχε υπηρεσίε ενδεχομένω παραβιάζουν του κοινωτικού κανόνε. Και ιστοσελίδε. Ε, παραπέμφθηκαν. Δηλαδή ε, ε, απευθυνθήκαμε στο κλάδο για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διδάσκεται από τις εμπειρίες αυτές και προετοιμάζει μια ανακοίνωση για την εφαρμογή του κεκτημένου ε, των καταναλωτών. Έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο και η ανακοίνωση αυτή θα κάνει μια απογραφή των δράσεων που έχουν ήδη αναλυφθεί και αν χρειαστεί θα αντιμετωπίσει οποιασδήποτε αδυναμίες και ελλείμματα για να ε, επιβάλλεται καλύτερα αυτό το δίκαιο των καταναλωτών. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι το θέμα της αποζημίωσης των καταναλωτών. Έχουν βέβαια δικαίωμα στην αποζημίωση όταν θίγονται από αθέμητες και παράνομες πρακτικές. Στην πράξη είναι πολλά τα εμπόδια για να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Ο κύριος λόγος αποτρεπτικός είναι το υψηλό κόστος. Ε, είναι η διαδικασία αυτή περίπλοκη της διένεξης εμπορικής. Δηλαδή ένας στους πέντε καταναλωτές ε, δεν προσφεύγει στα δικαστήρια για αξιώσεις κάτω των χιλίων ευρώ. Επιπλέον, οι καταναλωτές πολύ συχνά δεν γνωρίζουν ε, τι μέσα προσφυγής ε, διαθέτουν. Όλο και περισσότερο για πολλοί καταναλωτές, συγγνώμη, απογοητεύονται και δεν προσφεύγουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει το θέμα αυτό. Έχουμε παραγγείλει μελέτες, το έχουμε συζητήσει με τους ενδιαφερομένους και στο διαδίκτυο και πρόσφατα δημοσιεύσαμε μια πράσινη βίβλο όπου λάβαμε πάνω από 200 απαντήσεις. Παρόλο που τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς τρόπους προσφυγής, παντού υπάρχουν αδυναμίες. Υπάρχουν ε, ε, θέματα που είναι η και η που είναι εναλλακτικέ μορφές επίλυση διαφορών, αυτά υπάρχουν σε κάποια κρατημέλια, αλλά όχι σε όλα. Μόνο σε 13 κρατημέλη υπάρχει το δικαίωμα της συλλογική αγωγής. Αλλά και εκεί που υπάρχει, τα τελευταία χρόνια, πολύ λίγε είναι περιπτώσει που έχει χρηστεί. Γενικά υπάρχει χώρο για βελτίωση του συστήματο αποζημίωση ή δικαίωση των καταναλωτών. Γι' αυτό Έχουμε εξετάσει πάρα πολλές ε, προτάσεις εναλλακτικέ με την πράσινη βίβλο, με εργαλεία δεσμευτικά ή μη για δικαστική οδό ή εξοδικαστική. Και η συνδυασμό και των δύο. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες τώρα, ε, απλώς θα σας πω ότι ε, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τα επόμενα βήματα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όποιο δρόμο αποφασίσουμε να λάβουμε έχουμε τώρα την ευκαιρία να κάνουμε αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας και της υποστήριξής μας και ε, σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς το συμφέρον των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη και πιο γρήγορη, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έξι από τα καλύτερα μέλη της Επιτροπής μας είναι παρόντα. Ε, δυστυχώς πολλοί είναι απόντες γιατί έχουν επιστρέψει στις χώρες τους λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Έχουμε όμως έξι πολύ δραστήρια μέλη εδώ μαζί μας, τα οποία φαντάζομαι θα παρέμβουν. Ο κ. Τουμπό, ο κ. Χάρμπορ, ο κ. Λέχτερ, Σβάμπ, Χέτ και Ρούλερ. Ακόμα ένας είναι τακτικά μέλη και δραστήρια πάνω απ' όλα. Φαντάζομαι θα θέλουν να παρέμβουν στην ε, συζήτηση. Έχουμε και εκπροσώπους όμως των Εθνικών Κοινοβουλίων. Λοιπόν, πρώτα θα δώσω το λόγο στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ακούσω πρώτα δύο εθνικούς βουλευτές και συνεχεία θα δίνω το λόγο και ένα Ευρωβουλευτή. Πρώτος, Φαρούτσα από τη Μάλτα. Έχετε το λόγο. Κύριε Φαρούτσα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτή την Επιτροπή για το θέμα του κανονικού δικαίου. Ειδικά μετά το γεγονός ότι στη χώρα μου, στη, Μάλτα, χιλιάδες ε, πολιτών ε, πλημμύρισαν τα γραφεία του κόμματος για να υπογράψουν κείμενα ζητώντας την διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών κατά της κυβέρνησης για την επιστροφή του ΦΠΑ που είχε πληρωθεί παράνομα για τέλη κυκλοφορία όταν αγόρασαν το αυτοκίνητό του στη Μάλτα μεταξύ του Μαρτίου 2004 μέχρι το τέλος του 2008. Ε, και αυτό μετά μια θετική απάντηση από τον, τον Επίτροπο Κόβαξ τον περασμένο Ιανουάριο προς τον συνάδελφό που κάθεται δίπλα μου, τον κύριο Λούις Γκρέκ, που είναι Μαλτέζος ε, Ευρωβουλευτής, όταν υπέβαλε μια ερώτηση για αυτό το θέμα. Η εθνικιστική κυβέρνηση ε, στη Μάλτα δεν ήθελε να συμμορφωθεί παρά την κατακραυγή αυτών των ε, καταναλωτών που επί χρόνια ήταν ανενημέρωτοι για τα δικαιώματά τους και επομένως δεν μπορούσαν να ζητήσουν και αποζημίωση. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Γκρέκ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και συμφωνώ ότι ο μόνος τρόπος που ο μέσος καταναλωτής μπορεί να προστατευτεί εναντίον της ε, έπαρσης της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ένα σύστημα όπου τα ιδιωτικά και κυβερνητικά συμφέροντα συγχωνεύονται σε ένα χωριστό και ανεξάρτητο σώμα που αποτελείται από διάφορα άτομα και μόνο αυτός ο φορέας θα μπορεί να αυξάνει και να ρυθμίζει τις τιμές σε αγαθά ειδικά, και υπηρεσίες βέβαια, ειδικά σε υπηρεσίες όπως η ΔΕΚΟ, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή τιμές για την αποχέτευση και φόρη του αεροδρομίου κτλ. Προκειμένου να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι και αποτελεσματικό και σύμμορφο με το δίκαιο σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα είχαμε αστρονομικές αυξήσεις στη τιμή της ενέργειας ε, στη Μάλτα ε, σε αδικαιολόγητα επίπεδα από την κυβέρνηση. Μόνο έτσι ο καταναλωτής, ο απλός πολίτης ε, μπορεί να προστατευτεί και να μην είναι θύμα κάποιων μαθηματικών τύπων ε, που αυξάνουν τους φόρους και τις τιμές μόνο και μόνο για να υπάρξει αύξηση των εσόδων ε, στα ταμεία τα κρατικά. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα προστασίας του καταναλωτή. Ακούσατε την περίπτωση της Μάλτας για το ΦΠΑ η ενημέρωση για τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές τους δίνει το δικαίωμα να αναζητήσουν αποζημίωση για αυτά τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του ΦΠΑ. Ε, η αποπληρωμή, η επιστροφή των ποσών αυτών θα γίνει τέσσερα χρόνια μετά, στην καλύτερη περίπτωση. Η κυβέρνηση ποτέ δεν αισθάνθηκε υποχρεωμένη να ενημερώσει το κοινό για αυτή την κατάσταση, που συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια. Η έλλειψη ενημέρωση στη Μάλτα οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Και αν δεν υπήρχε ο κύριος Λούις Γκρέκ και οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι έγραψαν ε, προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, ε, θα είχαν παραμείνει αδαείς, ανενημέρωτοι οι καταναλωτές και θα είχαν μείνει στο έλεος της κυβέρνησης θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του καταναλωτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, να δούμε τι πρέπει να γίνει και να έχουμε άμεσα εφαρμοστικά μέτρα, ακόμα και κατά των κυβερνήσεων, ε, ειδικά όταν αυτές δεν συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τους καταναλωτές. Ακόμα... Θα ακούσουμε την επόμενη παρέμβαση και μετά ξανά τις ε, ευρωβουλευτές. Παρακαλώ να περιοριστείτε στα τρία λεπτά όμως για να μπορέσουμε να μιλήσουν όλοι. Κυρία Καλαμαλία από την Γαλλία. Σε μικρόφωνο ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, δώσατε κάποιες απαντήσεις στην παρέμβασή σας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των καταναλωτών. Γι' αυτό ακριβώς ε, υποστηρίζουμε την, την πρόταση οδηγίας. Έχουμε την αίσθηση ότι όλες ε, οι επιπτώσεις αυτών των φιλόδοξων επιλογών για μια μέγιστη εναρμόνιση για το θέμα αυτό δεν έχουν προσμετρηθεί σωστά. Γι' αυτό ακριβώς ε, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών θεωρούν ότι το κείμενο ευνοεί τι επιχειρήσει και όχι τους καταναλωτέ. Είπατε, το είπατε και στην αρχή της ε, παρέμβασής σας. Συμφωνούμε με αυτό το αίσθημα των καταναλωτών, γιατί πολλά από τα ερωτηματικά μας μένουν αναπάντητα. Επομένως είναι σημαντικό να αρθούν οι αμφισημίες, γιατί ο στόχος ε, για το μέλλον είναι να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός κώδικας για τους καταναλωτές. Επομένω, μια αμφιβολία είναι το πεδίο εφαρμογής ε, που ποικίλει από άρθρο σε άρθρο και κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Αυτέ οι εξαιρεσει δεν έχουν την ίδια εμβέλεια επίση σε περιπτώσει. περιπτώσεις. Ε, και μερικέ φορέ οι εθνικέ διατάξει παρεμβαίνουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν ισχύουν εθνικές διατάξεις. Επίσης, ε, υπάρχει ένας υπερβολικός φορμαλισμός. αφορά και τα κοινά καταναλωτικά αγαθά, όπω το ψωμί ή εφημερίδες. Επίση, ποια είναι η σχέση, ποια είναι η διάρθρωση με το αστικό δίκαιο. Στη Γαλλία ε, υπάρχει μια ανησυχία για την ικανότητα να συνεχίσουμε τις ίδιες εγγύησεις ε, και τα ίδια προβλήματα και να συνεχιστούν τα ίδια προβλήματα που είναι κρυμμένα στον αστικό κώδικα. Μας επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, τι γίνεται με τις καταχρηστικές ρήτρε και με το μηχανισμό και αν εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός, τότε υπάρχει μείωση του επίπεδου προστασίας. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί θεμητό αν δημιουργεί τέτοιες οπισθοχωρήσεις λόγω των καταχρηστικών ρητρών. Θέλουμε και διορθώσει από την Κομισιόν και ε, διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Uh, ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε ένα συνάδελφο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Χάρμπορ, συντονιστή του ΕΛΚ για την ε, Επιτροπή μας. ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμά του συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις για την σημασία όπως εμείς ε, θεωρούμε για την αυξημένη μπλοκή μας στον τομέα αυτόν, γιατί πραγματικά συνειδητοποιούμε ότι το πώς εφαρμόζεται επιτόπου το δίκαιο του καταναλωτή, το πώς αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα του καταναλωτή και οι μηχανισμοί των κρατών μελών αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του δικαίου στο ευρωπαϊκό επίπεδο και οπωσδήποτε είναι ευρύτατε οι διαβουλεύσει, αλλά εσεί όλοι είστε αιρετοί εκπρόσωποι και θα συνεργαστούμε και με τι αρχές σας και με τις ε, κυβερνήσεις σας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Παραγγείλαμε πρόσφατα μία μελέτη για τη μεταφορά επιτόπου της οδηγίας περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών, όπου είχαμε πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Γενικά νομίζω πως ήταν σημαντική πρόοδος, αυτή την εντύπωση έχουμε, αλλά μπορεί να έχετε διαφορετικές απόψεις βεβαίω, αλλά ναι, εδώ πέρα έρχομαι στο βασικό μου επιχείρημα στη ε, περιγραφή, κυρία Πρόεδρε, του έργου μας. Εάν ε, σκεφτείτε πως εξετάζουμε τη στρατηγική και το σκεπτικό των πραγμάτων και αμφισβητούμε κάποιες από τις υποθέσεις, αλλά προσπαθούμε να δούμε και το πώς θα προχωρήσει αυτή η πρόταση, έχουμε μια ιδανική ευκαιρία για να εμπλακείτε και εσείς ε, σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα αυτό γίνεται ήδη στη Βουλή των Λόρνων στη χώρα μου, αλλά για πρώτη φορά νομίζω τα τελευταία χρόνια μπορείτε να εμπλακείτε όλοι σε μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς ε, θα προχωρήσει η διαδικασία και εγώ συγκεκριμένα θα ήθελα να επισημάνω εδώ την πρόταση, την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων της Κομισιόν που για εμάς αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι των ε, ερευνών μας και θέλουμε να ακούσουμε πώς τη βλέπετε εσείς γιατί από εκεί θα οδηγηθούμε στα πλεονεκτήματα της μέγιστης εναρμόνισης. Ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα επιτόπου και ποια είναι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν για τους καταναλωτές της χώρας σας. Και αν ε, πραγματικά υπάρχει αύξηση των ωφέλους για το διασυναριακό εμπόριο, γιατί αυτή είναι η ισορροπία που πρέπει να βρούμε. Και πράγματι εμείς θέλουμε να προχωρήσει η εσωτερική αγορά, αλλά οπωσδήποτε όχι εις βάρος ε, τον ε, του αισθήματο προστασίας των καταναλωτών που θα πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα προστασίας και θα πρέπει να ξέρουν πού να απευθυνθούν για τυχόν ε, επανορθώσεις. Οπότε είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συνεδρίαση. Βεβαίω εμεί έχουμε ευρωεκλογέ, αλλά θα μπορούσατε ίσω κάποια στιγμή να επανέλθετε με τι προτάσεις Σα Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρένστρεμ τώρα από την Σουηδία. Fru ordförande, allmänt sett är Sverige till förslaget och Ευχαριστώ. Η Σουηδία είναι θετική απέναντι σε αυτήν την πρόταση γενικώ πώ. Υποστηρίζει επίση την πλήρη εναρμόνιση. Ούτω ώστε να έχουμε ένα σοβαρό επίπεδο προστασία του καταναλωτή. Η πλήρη εναρμόνιση μα δίνει αυτή την προστασία και βασίζεται σε νομικέ διατάξει ε, για την προστασία του καταναλωτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι επαρκή η προστασία του καταναλωτή και δεν θα, δεν θα θέλαμε να κινηθούμε προς την ε, λανθασμένη κατεύθυνση. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρξει εναρμόνιση προς τα κάτω. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εναρμόνιση για να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι θα βελτιώσουμε έτσι την κατάσταση των καταναλωτών αλλά και των εμπορευμένων και θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στο διασυνοριακό εμπόριο. Πιστεύουμε ότι έτσι θα υπάρξει περισσότερο ανταγωνισμό και επομένω και καλύτερε τιμέ, φθηνότερε τιμέ. Ε, φαντάζομαι ότι το επίπεδο προστασία του καταναλωτή θα κρατηθεί ψηλά. Αυτό είναι προ όφελο και των καταναλωτών και των εμπόρων. Η οδηγία έχει κάποιε διατάξει που πιστεύουμε ότι είναι ασαφείς. Παραδείγματο χάρη, εξετάσαμε την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και είναι πολύ σημαντικό το κείμενο να διατυπώνεται με ένα τέτοιο τρόπο που τα δύσκολα θέματα να είναι εύληπτα, γιατί είναι σημαντικό να τα καταλαβαίνουν και οι καταναλωτέ και οι έμποροι. Θα πρέπει οι κανόνες όχι μόνο να είναι αρμονισμένοι, αλλά και ξεκάθαροι και προβλέψιμοι. Πιστεύω ότι οι κοινοί κανόνες θα μπορούσαν να αυξήσουν σε μια αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων και αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου. Ευχαριστώ. Κύριε Κούνεγκεν, από τη Σλοβενία. Μπορεί βέβαια να μην προφράσω το όνομά σας, αλλά μπορείτε να με διορθώσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ όλους τους συναδέλφους, εξ ονόματος των Σλοβαίνων συναδέλφων. Νομίζω ότι ένας γενικός συντονισμός δεν θα πρέπει να υποσκάψει το υψηλό επίπεδο προστασίας ε, ε, των καταναλωτών όπως υπάρχει σε ε, ορισμένες χώρες, Φερρυπίν στη δική μου. Επί πολλά χρόνια προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, κάναμε πάρα πολλή δουλειά και αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια μείωση της προστασίας των καταναλωτών, σε μια πορεία προς τα κάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Προφανώς έχουμε ε, κάποιες επιφυλάξεις, κάποιες αντιρρήσεις, Η δική μας μόνιμη αντιπροσωπεία έχει εκφράσει τις, αντιρρήσει τις αντιρρήσεις ε, της Σλοβενίας. Αλλά πιστεύουμε ένα βασικό στοιχείο είναι να ενσωματώσουμε και τις ε, δημόσιες εταιρείες. Νερό, ε, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα. Και επιπλέον θα πρέπει να διευκρινίσουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις ε, που έχει, θα πρέπει να δούμε και τι καθήκοντα και τι δικαιώματα έχει. Όταν υπάρχει απόσυρση από μία σύμβαση. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ε, τα έχουμε ήδη παρουσιάσει. Επίσης, στην οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μια εύληπτη ε, διατύπωση και θα πρέπει να είναι και διατυπωμένη στη γλώσσα των καταναλωτών. Επομένως, επίσης, σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Επίσης, ο καταναλωτής ή μάλλον η Σλοβενία θέλει να προστατεύσει και τους καταναλωτές ε, που ψωνίζουν στο ίντερνετ. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εμπορίου γίνεται στο ίντερνετ. Έχουμε διάφορες επιφυλάξεις για το τέταρτο κεφάλαιο της πρότασης. Επίσης υπάρχουν τμήματα της οδηγίας όπου νομίζω ότι υπάρχουν λάθη, έχουν παρισφρήσει λάθη που μας οδηγούν σε μείωση της προστασίας του καταναλωτή. Κάτι που δεν είναι επιθυμητό βέβαια. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά είδη προσφυγής. Παραδείγματο χάρη μπορεί να επιστρέψει το εμπόρευμα ή να έχει άλλα μέτρα προσφυγής. Ε, η πρόταση οδηγίας δεν ιεραρχεί αυτά τα μέτρα. Και ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα επιλογής. Συγγνώμη, υπάρχει, υπάρχει μάλλον μια ιεραρχία και πρέπει να τη σεβαστεί ο καταναλωτής, επομένως δεν έχει δικαίωμα επιλογής. Επίσης, για τις εγγύησεις. Πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση, όχι να την αναρμονίσουμε πάση θυσία. Πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα, ιδίως σε περίοδο κρίσης. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων πρέπει να εξασφαλιστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή κατάσταση για όλους. Ο κ. Τουμπών τώρα. Από την Ευρωβουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα λίγο να πω Κάτι σχετικό με αυτό που είπε προηγουμένω ο κύριο Χάρμπορ. Θα ήθελα καταρχήν να αποτύσω ένα φοροτιμή στην πρόεδρο μα και στην επίτροπό μα, γιατί και οι δύο έχουν αφιερώσει πολύ μεγάλη ενέργεια εδώ και φαντασία. Και θα μας χρειαστεί αυτό για το μέλλον. Όταν θα ζητήσουμε την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν είναι ένα τομέα σίγουρα ε, στον οποίο μπορούν να γίνουν βήματα αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Βεβαίω είναι εξόχως πολιτικό το ζήτημα. Σχόλιο δεύτερο. Αρχίσαμε συζητάμε και είδαμε ότι ε, η πρόταση έχει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, αυτό της μέγιστης εναρμόνισης, ξέρετε. Και σήμερα η συγγήτριά μας, η κυρία Μακάρθη, προετοιμάζει ένα έγγραφο το οποίο θα μας υποβάλει και θα είναι πάρα πολύ ανοιχτό, γιατί όπως είπε και ο Χάρμπορ δεν είχαμε το χρόνο να εξετάσουμε αυτό το θέμα σε βάθος. Θα σας έλεγα λοιπόν εδώ ότι εγώ ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Δύο-τρία πράγματα γνωρίζω, χωρίς να έχω διαμορφώσει τελική άποψη. Πρώτον, σε ένα κόσμο σαν το σημερινό, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως πρόφαση την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικής οικονομίας που έχει να αμφισβήτητη, δεν μπορεί λέγω να βασιστεί πάνω σε αυτό για να ε, διακυβευθούν στοιχεία αυτού που ονομάζουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, πρότυπο. Έχουμε την αίσθηση σήμερα λοιπόν ότι αν η Ευρώπη μπορεί να εμφανίζει κάποιες αντιστάσεις ακόμα απέναντι στην κρίση, είναι ακριβώς γιατί έχουμε σωρέψει, πώς να το πω, ε, ε πολλή νομοθεσία, πολύ ε, στοιχεία που είναι κοινωνικοί προφυλακτήρες, ασπίδες και πρέπει να το σκεφτούμε. Η εσωτερική αγορά καλή είναι, και η διασυνοριακή κατανάλωση και απαραίτητη και για την ανάπτυξή μας, αλλά προσοχή. Αυτό που είναι ατού και γεκτημένο να μην διακυβευτεί. Παρατήρηση δεύτερη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δώσει μελέτη ε, πάρα πολύ εμπεριστατωμένη των επιπτώσεων, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Να δούμε δηλαδή ποιε θα είναι οι επιπτώσει σε κάθε χώρο όταν έχουμε μέγιστη εναρμόνιση. Το είπε και ο Χάρμπουρ. Και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δεύτερον, τρίτον δηλαδή, γιατί το δεύτερο το είπα πριν. Η σημερινή συνεδρία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε εκπροσώπους εδώ των Εθνικών Κοινοβουλίων. Παρατηρώ ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια λαμβάνουν θέση αρνητική προσέξτε, απέναντι στην πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στο όνομα της επικουρικότητας. Η Άνω Βουλή στη Γερμανία, για παράδειγμα, Bundesrat, η δική μας γερουσία, που είναι το δεύτερο σώμα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ήδη δήλωσαν ότι η οδηγία αυτή είναι απαράδεκτη, διότι ε, διακυβεύει την αρχή της επικουρικότητας. Είμαι πεπισμένο ότι και η Βουλή των Λόρδων και η Βουλή των Κοινοτήτων ανάλογα θα αποφασίσουν στο προσεχές διάστημα. Και θα ήθελα να πω και στη Μαγδαλένα Κούνεβα ε, το εξή, Τη στιγμή που εμείς κυρώνουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, που τίνει να προστατεύσει περισσότερο την επικουρικότητα και τα ε, εθνικά κοινοβούλια είναι σαφές, προσέξτε το αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι εμείς παραμελούμε, ε, παραγνωρίζουμε την άποψη των ε, βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω και ακριβώς αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να την αφαιρέσουμε και στην εφαρμογή των κειμένων που έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι θαυμάσια και πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αυτή, διότι το κοινοβούλιο μας πολλά θα διδασκόταν από αυτή την εμπειρία. Όχι απλώς να ε, αποφασίζουμε κείμενα, να νομοθετούμε, αλλά βλέπουμε πώς εφαρμόζονται και τι συνέπειες έχουν στην πράξη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Um, Ευχαριστώ. Παίρνουμε συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, κύριο Κλόβα από την Τσεχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας για τη διοργάνωση αυτής της ε, συνεδρίασης και για το ότι επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε ένα τόσο σημαντικό σχέδιο οδηγίας που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επηρεάζει άμεσα τους ε, πολίτες μας. Σας δούμε τώρα την άποψη της ε, γερουσίας της ε, τσεχικής δημοκρατίας. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού δικαίου περί καταναλωτή, ξεκινώντας ήδη από την Περάσινη Βίβλο, το 2007. Αργότερα από το Υπουργικό Συμβούλιο Γερουσία απάντησε στα ερωτήματα της ε, Κομισιόν, στα ερωτήματα που είχαν τεθεί σε αυτή την πράσινη βίβλο. Και τότε είχαμε επισημάνει πως ε, ο στόχος ε, αυτός, δηλαδή η απλοποίηση της νομοθεσίας δεν θα επιτευχθεί εάν δεν ε, ορίσουμε ακριβώς ε, την Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία και τα υπόλοιπα νομοθετικά μέσα και χαίρομαι για το ότι η Κομισιόν έλαβε υπόψη το κοινό πλαίσιο αναφοράς κατά τη σύνταξη αυτής της ε, οδηγίας. Το σχέδιο οδηγίας απασχόλησε την γερουσία της ε, Τσεχίας στην ε, τελευταία της συνεδρίασης, της 26 Μαρτίου και στο ψήφισμά μας ε, υποστηρίξαμε την αρχή της πλήρους εναρμόνησης με στόχο να μειωθεί ο κατακαιρματισμός της νομοθεσίας και να υπάρχει πραγματική προστασία των καταναλωτών επίσης. Καλωσορίσαμε το ότι δίνεται έμφαση στην πληροφόρηση των καταναλωτών και όσον αφορά την νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρούμε πως κοινέ προδιαγραφές για την προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή πρέπει να βασίζονται σε, στον καταναλωτή τον ίδιο ο οποίος θα είναι ενημερωμένος και προσεκτικός. Μόνο έτσι μπορεί να λάβει μια σωστή απόφαση για το εάν θα κάνει όχι μια διασυνοριακή συναλλαγή. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ και σε εσάς και στο επόμενο Κοινοβούλιο καλή επιτυχία με αυτή την οδηγία και ελπίζουμε ο στόχος της ε, να επιτευχθεί. Δηλαδή θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και θα είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές και επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές. Σας ευχαριστώ, η κυρία Σόνιτσον από την Σουηδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε και ευχαριστώ την Επιτροπή για την εισαγωγή της. Πριν ε, γίνω βουλευτής, δούλεψα σε οργάνωση για, τις, ε, για την προστασία του καταναλωτή. Και εκεί με, συνάντησα προφανώς πολλά άτομα τα οποία επίσης ενδιαφέρονται για την προστασία του καταναλωτή. Στη Σουηδία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το επίπεδο προστασίας ε, των καταναλωτών. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, έκαναν πολλές προσπάθειες για αυτό το θέμα και είμαστε πολύ δραστήριοι. Όταν θέλουμε να εναρμονίσουμε λοιπόν ε, την προστασία του καταναλωτή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλαμε ε, να την εναρμονίσουμε προς τα πάνω, ούτω ώστε να μην μειώσουμε το επίπεδο προστασίας. Θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά την εμπιστοσύνη. Μπορεί να υποσκαθεί η εμπιστοσύνη αν αρχίζουμε τώρα να αλλάζουμε τους κανόνες. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που είναι πολύ καλές, αλλά με την πλήρη εναρμόνιση μπορεί αυτό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών να μειωθεί. Βεβαίω σε άλλα κράτη-μέλη μπορεί να αυξηθεί η προστασία. Εν πρέπει να δούμε αυτό το ισοζύγιο. Υπάρχουν ε, διάφοροι παράγοντε που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γλώσσα, ε, συστήματα πληρωμών, κοινωνική ασφάλιση, ε, παραδόσει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για του καταναλωτέ και να τα λάβουμε στα σοβαρά. Οι σοσιαλδημοκράτε θα ήθελαν να είναι ήσυχοι ότι η Σουηδία θα κρατήσει ψηλά το επίπεδο προστασία των καταναλωτών, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μα. Ευχαριστώ, κυρία Χέντ, που επίση είναι ε, Σουηδή, ε, ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής ε, αυτής. Και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τους ε, Σουηδούς ε, εθνικούς βουλευτές. Βασικά με κάλυψαν, γιατί και εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης από τη Σουηδία. Είμαι ικανοποιημένη που έχουμε την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα θέματα των καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία και η Επίτροπος Κυριακούνεβα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Χαίρομαι που είναι τόσο δραστήρια και συνεργάζεται τόσο πολύ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να έχουμε μια ανθούσα αγορά, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτέ είναι ικανοποιημένοι και έχουν εμπιστοσύνη σε αυτήν την αγορά. Γι' αυτό στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτέ έχουν την καλύτερη δυνατή προστασία. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, που εν πάση περιπτώσει κάτι αρχίζει να κινείται και οι σοσιαλδημοκράτες στο Κοινοβούλιο ε, χαίρονται πάρα πολύ ε, με τις προσπάθειες. Βέβαια πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Ε, πρέπει να βρούμε το χρόνο και όπως είπε και ο κύριος Χάρμπορ θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις οργανώσεις των καταναλωτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε την αρμόνιση, νομίζουμε ότι είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν θέλουμε να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας του καταναλωτή. Θέλουμε να έχουμε τον υψηλότερο δυνατό ε, κοινό παρανομαστή, την υψηλότερη δυνατή ε, προστασία. Μια και μιλάμε για την ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ίσως κάποιοι αρχίσουν να υποβλέπουν την προστασία των καταναλωτή. Παραδείγματο χάρη ο τραπεζικός τομέας. Θα πρέπει λοιπόν εμείς όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να μην ε, μειώσουμε το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή με τίποτα. Προχωράμε στον κύριο Βολουδάκη από την Ελλάδα. Ακουστικά παρακαλώ, με μικρόφωνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ε, ενδιαφέρουσα εισήγηση της ε, Επιτρόπου. Ε, είναι γεγονός ότι ο κατακαιρματισμός των εθνικών νομοθεσιών αλλά και η πολυπλοκότητα των τεσσάρων ενισχύει οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή είναι γεγονός ότι μπορεί να καταλήγουν ακόμα και σε αναποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και βέβαια και σε εμπόδια στο ε, διασυνοριακό εμπόριο. Γι' αυτό πολύ σωστά η Επιτροπή παίρνει την πρωτοβουλία να αναθεωρήσει την νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η πρόταση της οδηγίας ως έχει σήμερα ε, δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να αναπτυχθεί το διασυναλλογικό εμπόριο παρά στην ανάγκη της προστασίας του καταναλωτή. Δεν είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι τα ε, συμφέροντα καταναλωτών και επιχειρήσεων είναι αναγκαστικά ε, σε σύγκρουση. Αντιθέτω, πιστεύω ότι πρέπει να τα συνθέσουμε για να οδηγηθούμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερία και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα ε, μπορεί και να συγκλίνουν και πρέπει να συγκλίνουν τα συμφέροντα αυτά. Και ο καταναλωτή θα είναι ωφελημένο από την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και από την ανάπτυξη τη αγορά γενικά. Όμω η οδηγία ω έχει, ξαναλέω, η πρόταση και μάλιστα με τη διαδικασία της πλήρου αναρμόνιση, δεν είμαι πεπισμένο ότι θα ε, οδηγήσει στο άριστο αποτέλεσμα σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή. Στην Ελλάδα το 2007 η ελληνική κυβέρνηση ε, αναθεώρησε την νομοθεσία του καταναλωτή και έχουμε σήμερα ένα νόμο, πιστεύω, ε, πολύ αποτελεσματικό και ευρεία εφαρμογής ένα νόμο ο οποίος προβλέπει μία σειρά από καταχρηστικές πρακτικές, οι οποίες αν η πρόταση οδηγία υιοθετηθεί, θα πάψουν να θεωρούνται καταχρηστικές. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως ξέρετε, είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη, μια κυβέρνηση που πιστεύει στην αγορά, στην ελευθερία της αγοράς, όμως στην ελευθερία της αγοράς με κανόνες. Με κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν πρωτίστως τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ε, έχουμε λοιπόν μια σειρά από ε, καταχρηστικές πρακτικές που προβλέπονται σήμερα από την Εθνική Νομοθεσία ως καταχρηστικές, οι οποίες θα θέλαμε να παραμείνουν καταχρηστικές, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο καταναλωτής σε μια αγορά που διαρκώς διευρύνεται, διαρκώ αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, διαρκώ ε, αντιμετωπίζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, διαρκώ αντιμετωπίζει νέους αντισυμβαλωμένους, για τους οποίους δεν γνωρίζει πολλά, θα θέλαμε να διατηρηθεί η δυνατότητα ε, της χώρας να εφαρμόζει την ε, νομοθεσία αυτή. Και πιστεύω και όπως άκουσα και από άλλους ισχύει αυτό και για άλλες χώρες. Ε, πιστεύω ότι η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου θα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και για την διευκόλυνση της Ευρώπης να βγει από τις συνθήκες της ύφεσης, από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που όλοι ζούμε. Ε, δεν πρέπει όμως σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσουμε να διευκολύνουμε την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου περιορίζοντας το επίπεδο της προστασίας του καταναλωτή που σήμερα υπάρχει και σε επίπεδο ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο προς όφελος των καταναλωτών, είναι προς όφελος μακροπρόθεσμα και της αγοράς και του διασυνοριακού εμπορίου γιατί εάν οι καταναλωτές νιώσουν ότι το επίπεδο της προστασίας των δικαιωμάτων τους περιορίζεται, ότι το επίπεδο της προστασίας των δικαιωμάτων τους γίνεται, ε, είναι, είναι πια χαμηλότερο, τότε θα περιοριστεί και η εμπιστοσύνη τους ε, στην αγορά, άρα και η συμμετοχή του στην αγορά και αυτό θα είναι ε, το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους. Πιστεύω ότι μέσα από τη διαβούλευση αυτή θα πρέπει να προβούμε σε ορισμένες ουσιαστικές βελτιώσεις, ούτως ώστε να μην ε, καταλήξουμε σε χαμηλότερο επίπεδο προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη και να λύσουμε τα ορισμένα επιμέρου προβλήματα πολύ ειδικότερα όπω αυτά που ακούστηκαν γύρω από τι ημέρε ε, στι οποίε υπάρχει δικαίωμα επαναχώρηση στη μία χώρα ή ε, στην άλλη. Πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα, ειδικά μέσα στην περίοδο τη κρίση την οποία διερχόμαστε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον. Σα ευχαριστώ. Thank you. Um, and I have uh, Madame Mistrello Destro from Italy. Από την Ιταλία τώρα. Η κυρία Μιστρέλο Ντέστρο, παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Μας αρέσει η προσοχή που δίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όχι μόνο στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, στο να δούμε ποια είναι, ποιο είναι το επίπεδο εφαρμογής ε, των οδηγιών, αλλά και στη λήψη νέων πρωτοβουλειών για να ενδυναμώσουμε την προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό εν ώψη της μεγάλης ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης της Υπήρους μας. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επανεκκινηθεί η, σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και ε, επιχειρήσεων ειδικά σε δυνα... διασυνοριακές αγορές και μιλάω κυρίως και για αγορές μέσω ίντερνετ. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τέτοιες αγορές. Καταρχάς μπορεί κάποιος να βρει μια προσφορά ε, πολύ πιο ενδιαφέρουσα, πολύ πιο ευρεία. Μπορεί να μειωθούν τα κόστη των ε, ενδιάμεσων και να πετύχει καλύτερες τιμές. Από τις αναλύσεις που έχουμε των δεδομένων ε, προκύπτει ότι μπορούν αυτές οι αγορές να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αν εξαλειφθούν κάποια εμπόδια. Όμως, οι αγορές στο ίντερνετ ε, υπόκεινται σε πολλές απάτες και σε πολλές καταχρήσεις. Θα πρέπει καταρχάς να δούμε την κατάσταση του προϊόντος τη στιγμή της παράδοσης και να δούμε ε, τι γίνεται σε περίπτωση ελαττωμάτων, να μπορεί να επιστραφεί δηλαδή το προϊόν. Τη στιγμή που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η πρόταση, ε, ασχοληθήκαμε με αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη μέχρι στιγμής βασιζόμαστε σε μια ελάχιστη εναρμόνιση Απλώς κάποια κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα υπέρ του καταναλωτή. Η συνύπαρξη διαφορετικών ε, συστημάτων ε, εμποδίζει τις αγορές να δραστηριοποιηθούν σε περισσότερες εθνικές αγορές. Ε, εμποδίζει, συγγνώμη, τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε περισσότερες αγορές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, ούτως ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και εύκολη εφαρμογή των κανόνων και της οδηγίας με τρόπο μονοσήμαντο. Θα πρέπει να έχουμε μια δέσμη κανόνων ε, ε, εύληπτη, σαφή. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και μέσα ε, αποκατάστασης, αποζημίωσης, σαφή σε όλη την Ευρώπη. Ε, αναφέρομαι κυρίως και στο λεγόμενο class action, στην ομαδική προσφυγή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω στην Επίτροπο ότι το Κοινοβούλιο μας και η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή χαιρετίζει την Επίτροπο. Ξέρω ότι θα έρθετε στην Ιταλία στις 23 Απριλίου και επομένως ε, θα είμαστε σε θέση να τα ξαναπούμε με μεγάλη χαρά και φαντάζομαι θα επανέλθουμε και σε αυτά τα θέματα που είναι τόσο ενδιαφέροντα. Um, Ευχαριστώ. Ήρθε και η κυρία Ρόιτοβα που είναι μέλος ε, πλήρης της Επιτροπής Τακτικό και Αντιπρόεδρος και θα έρθει στη συνέχεια και ο κύριος Χάνσλιχ που είναι μέλος. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σφάπ, ε, Γερμανός Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τους συναδέλφους από τα Εθνικά Τινοβολία. Το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ γόνιμο ως διάλογο. Όποιος στην Ευρώπη ενδιαφέρεται και εργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα τέτοιο θέμα, έχει σε πρώτη φάση ε, μια πάρα πολύ υποκειμενική αντίληψη για τα δικαιώματα και την προστασία του καταναλωτού, ορμόμενος ο καθένας από τη χώρα του, από το δίκαιο και το πλαίσιο που επικρατεί εκεί. Βέβαια, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο καταναλωτής. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι ταυτόχρονα οι καταναλωτές είναι και εργαζόμενοι ή εργοδότες, επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς αυτό που μας απασχολεί πάντα στην Επιτροπή μας δεν είναι ποιον θα προστατεύσουμε περισσότερο, αλλά πώς θα έχουμε ένα καλό μείγμα, μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ενδιαφέροντων και των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Θα ήθελα δε εδώ να έρθω να προσθέσω ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να προστατεύεται με νομικά εμπόδια και φραγμούς τόσο υψηλούς για τους επιχειρηματίες, γιατί τελικά δεν θα μπορεί να αγοράζει τα προϊόντα που ψάχνει και θέλει ο καταναλωτής. Θα έχουμε στάση εμπορίου. πρέπει να είναι όσο ε, γίνεται ευρύτερη η επιλογή των αγαθών και των υπηρεσιών και των προϊόντων το επικυριακούνευα θα πρέπει να ξανασκεφτούμε μήπως η οδηγία αυτή μπορεί να συνεισφέρει και προς μια άλλη κατεύθυνση. Να πάρουμε μια απόσταση από την λεγόμενη μακδονάλντοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να λειτουργούν μόνο πολύ μεγάλες αλυσίδες με πάρα πολλά υποκαταστήματα και διγατρικες κρατη κράτη-μέλη κυριαρχούν στην αγορά ή μήπως ε, ε, θα πρέπει ακριβώ να στραφούμε προ το διασυνοριακό εμπόριο και το μικρό και το λιανικό και τους μικρομεσαίους. Αυτή είναι η ενιαία αγορά, όχι μεγάλες ή μόνο επιχειρήσει. Λοιπόν, αυτό που μου φαίνεται το πιο σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση είναι η ευρύτερη δυνατή επιλογή. Από την άλλη, θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές και να παραμείνει ψηλή εμπιστοσύνη τους στην προστασία που τους παρέχει το επίπεδο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, έτσι και αλλιώ ορισμένα πράγματα νομικά ακόμα εκκρεμούν. Ποιο είναι αρμόδιο για ποια νομικά συγκεκριμένα. Γι' αυτό, για να περάσει αυτό το νομοθέτημα, έτσι και αλλιώ θα πρέπει να υπάρξει πολύ στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Να προσέξουμε τώρα, να μην αρχίσουμε κάθε ξεχωριστό επίπεδο ε, προστασίας ε, στο κράτος μέλος μας να το έχουμε γνώμονα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο καθένας. Στόχος πρέπει να είναι ε, να έχουμε όλοι μαζί στο μυαλό μας τέλος τη συνολική εικόνα, τη συνολική αντίληψη και έννοια. Εξυπηρετεί αυτό τον Ευρωπαίο πολίτη, είναι προς όφελός του, είναι πλεονέκτημα, ακόμα και αν σε κάποια χώρα, σε κατώτερο επίπεδο υπάρχει ε, άλλη προστασία και αλλαγή προς τα πάνω προς τα κάτω. Τώρα βέβαια και προεκλογικά δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά θα παρακαλούσα η συζήτηση αυτή να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Όχι ο καθένας ε, ξέρω εγώ στο μέλλον να δρυμώ τι προστασία απολαμβάνει ο καταναλωτή, μου, αλλά οι 480 εκατομμύρια καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι προστασία έχουν συλλογικά. Ευχαριστώ και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση που θα ακολουθήσει. από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την οργάνωση αυτής της ε, συνεδρίασης και οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι πολύ σημαντικό για την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όχι μόνο να λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο η πολιτική των καταναλωτών αλλά και σε ευρωπαϊκό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις σχέσεις ε, μεταξύ του πολιτή και του πελάτη όσον αφορά τη σύμβαση, τη διαφήμιση μια υπηρεσία ή κάποιων αγαθών. Η ανάλυση δείχνει πως εάν υιοθετηθεί αυτή η νέα πρόταση μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία κάποιοι από τους ε, κινδύνους μετά από έξι μήνες θα μετατοπιστούν προς τον καταναλωτή και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Μήπως ε, δεν θα έπρεπε να αντικατοπτρίζουν τυχώς ε, προσεγγές τους όρους της σύμβασης. Επίσης, όταν μιλάμε για τους κατασκευαστές, καλό είναι να μην διαταράσουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων από την πλευρά των ε, καταναλωτών. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ασφάλεια και εμπιστοσύνη, αλλά και οι επιχειρήσεις από την ε, πλευρά τους πρέπει να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μέσω της ε, ποιότητας και τέλος το νομικό περιβάλλον όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Εγώ συμφωνώ με όσοι λένε ότι θα πρέπει να είναι απλό αυτό το και άρα κατανοητό από τους καταναλωτές. Ε, Αυτή πρέπει να είναι η προσδοκία από πλευράς ε, του καταναλωτή, αλλά βεβαίως το περιβάλλον αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, γιατί αυτό μεταφράζεται σε κόστος. Γιατί μετά το αποτέλεσμα στην ε, οικονομία είναι ότι θα ανέβουν οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο στην ε, σχέση καταναλωτή και επιχείρησης είναι η πληροφόρηση, η σωστή πληροφόρηση για τα αγαθά και τις ε, υπηρεσίες. Τελειώντας λοιπόν, θα ήθελα να υψημάνω πως η εποπτεία της αγοράς, η εισαγωγή νέων κανόνων και η αξιολόγηση των αντικτύπων τους θα πρέπει να γίνεται με βάση τα το ίδιο μέτρο και τότε μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί και με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Νομίζω πως αν ε, είναι ενιαία η ερμηνεία τα πράγματα θα είναι απλούστερα. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω το ότι χρειάζεται και η διαβούλευση ε, με τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ κύριο Στόντσεκ από την Αυστρία. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από τα Ευρωπαϊκά από τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι πρόεδρος της ίδιας επιτροπής στο Εθνικό Συμβούλιο της ε, Αυστρίας και οπωσδήποτε το σημαντικό αυτό ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών μας απασχολεί και σε εθνικό επίπεδο όπως και σε ευρωπαϊκό. Αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Υπόθεση στην οποία όλοι νομίζω σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει μία κοινή οδηγία που κάποια πράγματα θα τα εναρμονίσει, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προχωρήσουμε στην πλήρη εναρμόνιση γιατί θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε προς τα πάνω και όχι ε, προς τα κάτω. Και αν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση προς τα πάνω και ίσως κάποια πράγματα θα πρέπει να ε, εναρμονιστούν προς τα κάτω. Και εδώ πέρα είναι και το θέμα της νομολογίας, νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε στην ελάχιστη εναρμόνιση και να διατηρηθεί νομίζω η αρχή της ε, χώρας προέλευσης διθλάμβους να πάμε να παραπέρα και κυρίως ε, σε σχέση με αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα π.χ. σε τομείς όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης ή οι διαφορετικές προθεσμίες. Έχουμε... Αναφέρθηκε ήδη το πώς ε, μετράμε τις μέρες, αν εργάσιμες ή όχι. Εντάξει, ναι, αυτό να το εναρμονίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει συγκρισιμότητα, Κυρίω όταν μιλάμε για τιμέ ενέργεια ρεύμα, φυσικό αέριο, βενζίνη. Επίσης ε, να υπάρχει συγκρισιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων. Ε, δεν συμβαίνει αυτό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τα τέλη των αεροδρομίων και τα αεροπορικά εισιτήρια. Νομίζω ότι ε, με μικρά βήματα εδώ πέρα μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με πλήρη εναρμόνιση, γιατί θα έχουμε αρκετές δυσκολίες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλερ, που είναι συντονίστρια των Πρασίνων. Ευχαριστώ και εγώ χαιρετίζω αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ δεν έχω κατασταλάξει όσον αφορά την απόψή μου. Θεωρώ πως είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία της κυρίας Κούνεβα και είναι σημαντικό το ότι συστάθηκε στην Επιτροπή μας μια ομάδα εργασίας που θα δει το θέμα αυτό σε βάθος και θεωρώ πως η σημερινή ανταλλαγή απόψεων σήμερα μας βοηθά γιατί κυρίως τα προβλήματα είναι στη λεπτομέρεια. Για μένα λεπτομέρεια σημαίνει πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ακριβώς ειδικά όσον αφορά την αναλογικότητα, την επικουρικότητα, τι ακριβώς νόημα έχει η πλήρης εναρμόνιση και που, ε, τι είναι το καλύτερο να κάνουν τα, τα κράτη-μέλη Ίσως θα έπρεπε να μην ε, προχωρήσουμε στην πλήρη εναρμόνιση, να μείνουμε στην ελάχιστη εναρμόνιση. Βεβαίως η πλήρη εναρμόνιση έχει το εξή ε, πρόβλημα, ότι μετά δεν υπάρχει καμία ευελιξία στα κράτη-μέλη, δηλαδή το κράτος μέλος μετά δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει γρήγορα εάν αλλάξουν οι αγορές. Με την πλήρη ε, εναρμόνιση είναι αυτό το θέμα, αλλά βεβαίως μπορεί αυτό να αποβεί και θετικό. Θα, το, θα πρέπει να το δούμε αυτό σε βάθος και λοιπόν για το ότι η μελέτη αδικτύπου της Κομισιόν δεν μας δίνει ακριβώς πολλές λεπτομέρειες για το ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στα κράτη-μέλη για να το δούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θεωρώ πως εμείς ως ε, βουλευτές ε, ε, λάβαν πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτημα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ειδικά σε όλη αυτή την πρόταση και τελευταία παρατηρήση και δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με το πεδίο εφαρμογής γιατί θεωρώ πως ε, το έβρος αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και να συμπεριλάβουμε μόνο τμήματα της ε, ε, οδηγίας. Δεν ξέρω κατά πόσον θα περιοριστεί αυτός ο κατακαιρματισμός εάν μειώσουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, πω ότι συμφωνώ, έχουν δίκιο εκείνοι που λέγουν και τους υποστηρίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε ε, και προειδοποιούν για την πλήρη εναρμόνιση και τις επιπτώσεις της. Γιατί και εμείς στην Αυστρία έχουμε ήδη πολύ ψηλή ε, προστασία του καταναλωτού και φοβόμαστε ότι με την πλήρη εναρμόνιση αυτό θα μειωθεί δραστικά ή τουλάχιστον θα είναι διάτριτο στη συνέχεια το σύστημα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ελάχιστη εναρμόνιση. Γιατί ακριβώ δεν είναι πλήρη εναρμόνιση και δεν μπορούμε να διατηρήσουμε του πιο αυστηρούς κανόνε που ισχύουν στην Αυστρία. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλοι φόβοι και μεγάλες αντιστάσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι η σταδιακή ρύθμιση θα ήταν η ιδεώδης λύση με διαφοροποίηση της προσπάθειας, με ελάχιστη εναρμόνιση τουλάχιστον και σε τομείς πλήρη εναρμόνιση. Ιδιαίτερα για την εναρμόνιση του κειμένου δικαίου καταναλωτών. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε να μην χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση και επικρατήσει ε, ελεύθερη αγορά. Ε, ε ασίδατη δηλαδή. Επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε ελάχιστη εναρμόνιση. Στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει σε ορισμένε περιπτώσεις και μάλιστα προσφέρονται ορισμένε διατάξει και για πλήρη εναρμόνιση. Παράδειγμα, η πώληση εξ αποστάσεως. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες σαφείς, όπως είναι α πούμε οι στο διαδίκτυο, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις ε, για τα ε, συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες, εξαιρέσει τις υπηρεσίες. με προθεσμίες διάφορες για ανάκληση, για ε, καταγγελία της σύμβασης. Θα πρέπει ο καταναλωτής να γνωρίζει τα δικαιώματα του, το επιμηκύνεται η προθεσμία παρισυλλογής και μόνο δεν σημαίνει τίποτα. Και οποιασδήποτε θέμη τις πρακτικές θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά. Γενικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να στήσουμε τώρα έναν ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων και επιπέδων προστασίας στην αγορά και των συμφερόντων των καταναλωτών. Θα πρέπει μάλλον να ε, προσανατολισμούμε στο ποιο αξίζει περισσότερη προστασία, για ποιο είναι ο πιο δυνατό. Αυτό είναι σίγουρα ο καταναλωτής. Αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε και δεν θα πρέπει καθόλου να είμαστε φιδωλοί στι ε, αξιώσεις και στις απαιτήσει για την ποιότητα και για την ασφάλεια. Και αυτό θα ενισχυθεί και διεθνώς στις αγορές. Και ξέρουμε όταν υποχρεώνονται δια νόμου σε μια συμπεριφορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό δρά δημιουργικά. Τους ε, ε, παροτρύνει να προχωρήσουν σε καινοτομία, σε ανάπτυξη και έτσι υπάρχει και μεγάλη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των πολιτών μας. Και θέλουμε την Ευρώπη των πολιτών εμείς, όχι την Ευρώπη των ομίλων και των μεγάλων εταιριών. Το πιο αδύναμο πρέπει να προστατεύουμε στην αγορά. Ξέρω ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό. Και εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στην κυρία Επίτροπο, στην κυρία Κούνεβα, καλή επιτυχία για αυτό το δρόμο που θα είναι επίπονος. Ε, ε, Ευχαριστώ. Η κυρία Ολιβέηρα από την Πορτογαλία έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση που μας στείλατε και μας επιτρέπετε να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η οδηγία εκ των πραγμάτων είναι ένα σημαντικό βήμα για την ε, προστασία του καταναλωτή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά για να φτάσουμε στο σωστό σημείο ισορροπίας. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται όμως αυτή η οδηγία για να και για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και για να τον ενημερώσουμε. Θα ήθελα να σας πω κάτι συγκεκριμένο για την ε, επιβλαβή διαφήμιση, τόσο σε ό,τι αφορά τα αγαθά, όσο και τις υπηρεσίες. Συχνά οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας της διαφήμισης που τους ε, παραπλανά εντελώς. Αναφέρομαι κυρίως στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις διαφημίσεις που κάνουν. Έγιναν διαφημίσεις προϊόντων με τρόπο που πραγματικά μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή ή με τρόπο που εξαναγκάζει τον καταναλωτή να αγοράσει διάφορα προϊόντα. Ανησυχώ για αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει σε διάφορες χώρες και θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τι μπορούμε να κάνουμε εν συνεχεία και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Ποιοι είναι οι κατάλληλοι μηχανισμοί. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους τομείς να αποφύγουμε την συνεχή παραπλάνηση των καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ήρθαν. Ο κύριος Όσκαρς Κάστενς από τη Λετωνία, παρακαλώ. Συνεχίζουμε δηλαδή με τους εθνικούς βουλευτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, για την πρωτοβουλία αυτή για την ανταλλαγή απόψεων για το δίκαιο των ε, καταναλωτών. Βεβαίως ο πρώτος ε, σχετικός ε, νόμος ε, σε μας πέρασε το 1990 ήδη με βάση την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα υπάρχει το κέντρο προστασίας καταναλωτών αλλά και αρχές τομεακές τους διάφορους κλάδους. Όσον αφορά τώρα την οδηγία η οποία θα τεθεί ενισχύ όλα αυτά μεταφέρονται στο Εθνικό Δίκαιο με αποφάσεις του Υπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. Ε, εν πάση περιπτώσει εμείς ε, θα προτιμούσαμε ένα υψηλότερο επίπεδο και έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτά τα οποία προβλέπουν οι φυστάμενες οδηγίες, π.χ. όσον αφορά τις εξαποστάσεις πωλήσει μπορεί να υπάρξει επαναχώρηση εντός 14 ημερών χωρίς ε, καμία, κανένα πρόβλημα, ενώ η οδηγία προβλέπε 7 ημέρες. Εμείς ε, λοιπόν είμαστε υπέρ της μέγιστης ε, εναρμόνισης που προτείνεται στην οδηγία, αλλά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα νερώσουμε με αυτό το μέτρο τις υφιστάμενες προδιαγραφές. Η πείρα μας δείχνει πως ε, δεν ε, είναι πάντα δεν υπάρχει πάντα εγγύηση για το δικαίωμα του καταναλωτή στην ελεύθερη επιλογή. Κατά την άποψή μας η προσέγγιση της πλήρους εναρμόνισης όπως ε, δείχνει και η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, ε, εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε στο Κοινοβούλιο το τι θα μπορεί να γίνει με τις προσφυγές για την σήμανση των τροφίμων, καθώς είχαμε και παραπονά και προσφυγές των καταναλωτών και αφορά βεβαίως και την σχετική οδηγία για την ε, σήμανση των ε, τροφίμων. Γιατί συχνά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και είναι και πολύ μικροί οι χαρακτήρες της ε, ετικέτες, δεν αναγράφεται το εάν έχουμε γενετικά τροποιημένους οργανισμούς, οπότε παραβιάζεται το δικαίωμα πληροφόρηση του καταναλωτή για το εάν λάπτο πιθανώς στην υγεία του αυτά τα προϊόντα τα οποία θα καταναλώσει. Επίσης ε, μια άλλη εταιρεία έδινε πληροφορίες μόνο κατόπιν αιτήματος και αν ζητούσε μια απαραίτητη έκπτωση Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει εμείς θεωρούμε, για να κάτι άλλο, να, πως θα πρέπει να αναφέρεται και ο κατασκευαστής και η προέλευσή του, εάν είναι να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εναντίον του ο καταναλωτής. Ειδικά τώρα στην περίοδο κρίσης στην οποία βρισκόμαστε, η νομοθεσία για ομαδικές ε, πρόσφυγες, αλλά και για την ε, συλλογική ε, προστασία των καναλτών πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει επίσης όμως ταυτόχρονα να εισαχθούν και νωρίτερα μάλιστα οι μηχανισμοί εξοδικαστικής ε, επίλυσης ε, των διαφορών και μάλιστα να είναι προσβάσιμοι σε όλες τις χώρες, ειδικά όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών. Θεωρούμε επίσης πως το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών αυτή τη στιγμή στις υπάρχουσες οδηγίες δεν θα πρέπει να μειωθεί. Εμείς ε, θεωρούμε πως θα πρέπει η οδηγία να προσφέρει κάτι απτό για την ενίσχυση των δικαιωμάτων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ. Η κυρία από την... Ο κύριος Τουμπιτούλη, με συγχωρείτε Ε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Πιστεύω όντως ότι πρέπει να προχωρήσει το θέμα χωρίς καθυστέρηση η σημερινή οικονομική κρίση μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο την προστασία στα κράτη-μέλη. Ε, ειδικά τα μικρά κράτη με μικρότερες οικονομίες χρειάζονται ε, βοήθεια για να λειτουργήσει καλά ε, η αγορά τους και η κοινωτική αγορά εν γέννη. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό λοιπόν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Εμείς ε, συμφωνούμε με τις αρχές οδηγίας σε ό,τι αφορά το δίκαιο των καταναλωτών. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό εμπόριο, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων ε, στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν η μεγαλύτερη ομοιογένεια είναι σε συμφωνία με τους στόχους μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ε, όπως αυτές που είπαν και άλλα κράτη-μέλη, ιδίως η Σλοβενία και η Αυστρία. Οι επιφυλάξεις μας ε, αφορούν κυρίως τις διατάξεις για τις συμβάσεις ε, πωλήσεων. Εμείς έχουμε στην εθνική μας νομοθεσία τέτοιου τύπου διατάξεις και φοβάμαι ότι οι διατάξεις οδηγίας θα επηρεάσουν αρνητικά αυτού του είδους της πολίτης σε βασικούς τομείς, κυρίως το δικαίωμα υπαναχώρησης από το, τη σύμβαση και αντί για δύο χρόνια ευθύνη για τα ελαττωματικά αγαθά, ε, θα έχουμε εξαετή. Είχαμε εμεί στην εσωτερική μας νομοθεσία εξαετή περίοδο, αλλά αυτό αντικαθίσταται με τη διετή τώρα. Επίσης, Έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην εσωτερική νομοθεσία από την οδηγία για την παράδοση των αγαθών. Ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πλήρης εναρμόνιση με βάση την παρούσα πρόταση θα οδηγήσει σε προβλήματα στην Ιρλανδία. Σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους τομείς. Κύριος Πίτερ Χάουκ από τη Γερμανία. Βάτη Βιτεμβέργη πιο συγκεκριμένα, από τη Γερουσία της Γερμανίας. Κύριες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα περιγράψω σύντομα τη στάση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της Άνω Βουλής θα λέγαμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Επίτροπο για το σχέδιο οδηγίας που μας οδηγεί σε μια πολύ σημαντική συζήτηση και βεβαίως ε, μπορεί να αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά κατά το οποίο μας αφορά όλους στο πλαίσιο της στρατηγικής Λισαβόνας και το υποστηρίζουμε. Θεωρώ πως ε, σημαντικό είναι πραγματικά να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά πράγματι από πλευρά επιχειρηματικότητα, αυτό το οποίο αναφέρθηκε βεβαίω ω μακδοναλντοποίηση, αλλά να παραμείνουν ταυτόχρονα ζωντανέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ταυτόχρονα για τον καταναλωτή, για τον χρήστη, για τον πολίτη να ε, γίνει κάτι το ζωντανό ως χώρος ε, αγορών, ε, ταξιδιών, υπηρεσιών, διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο σπάνια. Η οδηγία, το σχέδιο αυτό οδηγίας έχει κάποια πράγματα στα οποία είμαστε επικριτικοί. Πρώτα απ' όλα είναι το περιορισμένο εύρος πεδίο εφαρμογής, δηλαδή αφορά τους γενικούς όρους των συμβάσεων στις εξαποστάσεως παροχής ε, πωλήσεων, υπηρεσιών κτλ. Θεωρούμε πως θα πρέπει να δημιουργηθούν πιο συνεκτικοί κανόνες ε, πλαίσιο για όλους ε, τους ε, τομείς συνολικά. Επίσης για εμάς όπως και για άλλα κράτη-μέλη θεωρούμε πως είναι σημαντική η πρόταση Κομισιόν να προτείνει πλήρη εναρμόνιση και νομίζω θα επιτύχουμε πλέον για την εσωτερική αγορά των καταναλωτών, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό να έχουμε πλήρη εναρμόνιση σε ορισμένους τομείς και αλλού να έχουμε μία ελάχιστη εναρμόνιση. Με αυτό τον τομέα βέβαια, με αυτή την ε, τακτική βεβαίως θα μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα αναλόγως με το τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Επίσης ε, αυτό το οποίο ανησυχεί τη Γερμανία είναι η μείωση του επίπεδου της ε, προστασίας των καταναλωτών. Επίσης έχουμε κάποιες αντιρρήσεις για τις λίστες αυτές τις γκρίζες και τις μαύρες. Καταρχήν ε, βεβαίως έχουμε ένα κάποιο επίπεδο ήδη στην ε, Γερμανία Προστασίας αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα θα καταρτίζονται στην επιτροπολογία όπου θα περάσουν και άλλες ρήτρες ε, και όλα αυτά θα θεθούν στη διακριτική ευχέρεια της ε, Κομισιόν και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία νομίζω θα πρέπει να παραμείνει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Επίσης έχουμε επισημάνει κάποια πράγματα στα οποία πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Θεωρούμε πως ε, στο μελλοντικό δίκαιο το ευρωπαϊκό του καναλτή θα πρέπει να έχουμε ένα εγγυημένο υψηλό επίπεδο ε, προστασίας που θα μας δώσει τη δυνατότητα και στο μέλλον να ανταποκριθούμε στις ε, πολιτικές ε, προκλήσεις αρκετά ευέλικτα. Σας ευχαριστώ. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η Βερόνι Χόρθ που είναι πρόεδρος υπό Επιτροπής της Βουλής των Λόρδων και βεβαίως εμείς ως Βρετανοί έχουμε πάντα επαφές με τη Βουλή των Λόρδων. Είμαι πολύ σύντομη. Η Βουλή των Λόρδων θέλει να κάνει μια πλήρη έρευνα ε, στην οδηγία. Είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Αυτό που μου άρεσε σήμερα το απόγευμα είναι ότι άκουσα τις ανησυχίες των άλλων κρατών μελών. Θα ήθελα όμως να διορθώσω κάτι που υπόθηκε πριν για την επικουρικότητα. Γιατί η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι θα υπάρξουν ωφέλη από την οδηγία. Για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενθαρρύνει η οδηγία αυτή την πλήρη εναρμόνιση, αλλά όχι ε, βάσει της σημερινή οδηγίας. Όπως είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι, υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στην ε, οδηγία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η κυβέρνησή μας πιστεύει, από μια πρώτη ματιά που κάναμε και στη δική μου επιτροπή, ότι αν προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μάλλον θα μειώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα την αυξήσουμε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, οι νομικές επιπτώσεις της οδηγίας, και βέβαια θα μάθουμε κι άλλα καθώς ε, μελετάμε το θέμα, θα είναι πολύ περίπλοκες. Θα πρέπει να απλουστευθούν, θα πρέπει να χτενιστούν όλα αυτά τα θέματα. Μια πρώτη γνώμη σας λέω. Ε, χρήσιμο θα ήταν αυτό το κείμενο, αντί να είναι οδηγία, να είναι μια λευκή βίβλος. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται. Οι καταναλωτές ε, θέλουν να, το οποιοδήποτε κείμενο να καλύπτει και τα αγαθά και τις υπηρεσίες, γιατί τους ενδιαφέρουν και τα δύο. Ελπίζουμε ότι και ο κλάδος και οι οργανώσεις των καταναλωτών και οι δικηγόροι θα μας ε, δώσουν τις απόψεις τους και αυτό θα μας βοηθήσει. Τα δύο βασικά σχόλια που θέλω να κάνω είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει για να υπάρξει μια κοινή κατεύθυνση, μια κοινή οδηγία. Η σημερινή κατάσταση, η σημερινή οδηγία θα είναι απαράδεκτη για τα κράτη-μέλη αν αυτή μειώσει την προστασία των καταναλωτών. Ε, και αποκλείεται να περάσει το κοινοβούλιο μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κρατήσει ψηλά την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών. κυρία Αλέξα από την Ουγγαρία. Κύριος, για την ακριβία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Ουγγρική Βουλή σας καλωσορίζει και εγώ εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς στην Ουγγρική Βουλή. Τα τελευταία χρόνια κάναμε πάρα πολύ σημαντική δουλειά για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ουγγαρία και στο έργο μας αυτό μας βοήθησαν και ε, τα νομοθετικά βήματα που έκανε ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, μπορώ να πω το εξής ως προς τη μεταφορά και την εφαρμογή του νόμου αυτού στην Ουγγαρία. Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση του έτους 1997, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά Και δεν έχει περάσει και πάρα πολύ χρόνος από, τότε, ε, από το νέο σύστημα δηλαδή και δεν μπορώ να σας ε, αναφέρω και λεπτομέρειες. Αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς και συγκεκριμένοι στην εφαρμογή και η πολιτική ε, με ομικρογιώτα, η κοινωνία των πολιτών και οι διάφορες άλλες οργανώσεις, σωματεία και σύλλογοι είναι ικανοποιημένοι με την παρούσα κατάσταση. Έχουμε κάνει τους κανόνες πιο αυστηρούς, τους έχουμε ενημερώσει, επικυρωπήσει και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Η Ουγγαρία υποστηρίζει αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ε, έννοια και την ε, εναρμόνιση προς τα πάνω. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ακριβείς ρυθμίσεις ε, σαφείς για να μην κάνει ο καθένας από εκεί πέρα τις δικές του ερμηνείες. Και όταν κάποιος έχει πιο αυστηρούς κανόνες ε, και πιο ε, ψύχρονη νομοθεσία δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Κοιτάξτε, πριν παραδώσω στην κυρία Ρόιτοβα την Προεδρία για τη δεύτερη συνεδρία που θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχουμε κεντρικού ομιλητέ. Εχθές είχαμε ένα μικρό εργαστήρι για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της μεταφοράς και της εφαρμογής. Θα ήθελα ε, να απαντήσει αν έχει την καλοσύνη η Επιτροπός, όχι στο καθένα ξεχωριστά προφανώς, αλλά σε μια γενική δευτερομιλία. Να δευτερολογήσει, να απαντήσει και Βεβαίω, αν συμφωνείτε, συμφωνείτε και εμεί συμφωνούμε με το ότι είναι σημαντικό αυτό ως νομοθεσία, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι η χώρα τους κάνει καλύτερα τα πράγματα στην προστασία. Δηλαδή όλοι είμαστε υπέρ, αλλά μερικοί είμαστε υπέρ της εθνικής μας νομοθεσίας περισσότερο από της κοινοτικής. Μα γι' αυτό κάνουμε προτάσεις, για να προσπαθήσουμε να λύσουμε και να βρούμε τη σωστή ισορροπία στη νομοθεσία. Η Επίτροπος έχει το λόγο και μετά ο κύριο Τζίλικ θέλει να πει μερικά πράγματα. Ζητώ συγγνώμη πρέπει να σα αφήσω, γιατί έχω άλλη ανηλυμένη υποχρέωση. Σα ευχαριστώ. Uh, Πολύ ενδιαφέρουσα όσα μα είπατε. Όλοι σα. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις προσδοκίες που έχω. πίστευα ότι θα ακούσω πολλές χώρες να λένε ότι η δική τους εθνική προστασία είναι καλύτερη από την κοινοτική. Είμαστε πεπισμένοι ότι όχι μόνο η Δανία και η Σουηδία που έχουν τις παλιότερες ε, οργανώσεις καταναλωτών θεωρούν ότι είναι πρωταθλητές της προστασίας, αλλά βλέπω και ότι η Πορτογαλία και η Ελλάδα θεωρούν ότι τα πάνε πολύ καλά. Είμαστε περήφανοι λοιπόν που βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια υπάρχει καλή προστασία, σε όλες τις χώρες. Καλό είναι αυτό. Γι' αυτό όμως χρειάζεται να έχουμε και μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί σε αυτό τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν αρκεί να τα πάμε καλά στη δική μας χώρα. Για να δούμε τι πιστεύει η Ευρώπη για την προστασία των καταναλωτών. Θα ήθελα να σας πω για ε, διαπραγματεύσεις που ε, έχω διενεργήσει με την Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν εκεί διαπραγματεύομαι, τους λέω τι πιστεύει η Ευρώπη. Προσπαθώ όχι να πουλήσω το patchwork από τις 27 κατακαιρματισμένες εθνικές νομοθεσίες, γιατί ναι μεν κάποιοι από εσά ε, είσαστε πάρα πολύ καλοί στις χώρες σας, τα πάτε πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ προσπαθώ να πείσω τους ξένους ότι η Ευρώπη είναι γενικά σε πολύ καλό επίπεδο. Και διαπραγματεύομαι ως επίτροπος υπεύθυνο για την προστασία των καταναλωτών. Ε, θέλω να υπερασπιστώ την Ευρώπη. Μιλάμε συνέχεια για την παγκοσμιοποίηση. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι για να προστατευόμαστε καλά ως καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αρκεί η εθνική νομοθεσία που είναι απλώς η αφετηρία. Έρχομαι σε επαφή με πολλούς Βρετανούς πολίτες, ακόμη και εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουν ανοιχτό πνεύμα. Θέλουν να δουν ποιε είναι οι πραγματικότητε. Θέλουν να προστατεύονται όχι μόνο στην Ομένη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα που πηγαίνουν για ε, Διακοπέ, Γι' αυτό έχουμε την οδηγία για τη χρονομενιστική μίσθωση. Ακόμη και αν κάποιο κάθεται στο σπίτι και απλώς παίζει με το ποντίκι του στον υπολογιστή. Ακόμα και έτσι μπορεί κανείς να επωφελείται από την εσωτερική αγορά. Λοιπόν, ξεκινήστε από αυτό. Έχουμε ένα διασυνοριακό εμπόριο που είναι, ε, έχει φτάσει στο ποσοστό του 6%. Όταν ξεκινήσαμε με το ευρωβαρόμετρο να ρωτάμε τους καταναλωτές γιατί δεν διερευνούν άλλες αγορές. Η απάντηση ήταν όχι η γλώσσα, εμεί αυτό νομίζαμε. Αλλά οι τελείω διαφορετικοί κανόνε, του οποίου δεν καταλαβαίνουν σε άλλε χώρε, δηλαδή αν πάνε στην Ισπανία ή στην Ελλάδα για διακοπέ, ή ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κανόνε δεν είναι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι με τη χώρα του ή αν θέλουν να αγοράσουν μια τηλεόραση στο εξωτερικό. Αν δείτε τις τιμές, έχουμε όλο και περισσότερα παρατηρητήρια τιμών. Βλέπετε ότι πρέπει κάποιος να κάνει μια προσπάθεια για να συγκρίνει τις τιμές. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν εμείς οι καταναλωτές να αισθανθούν ε, εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε τις επιχειρήσεις. Το 50% των επιχειρήσεων πουλάνε online, μέσα στη χώρα τους. Και αυτέ οι επιχειρήσει, το 50% των επιχειρήσεων, θέλουν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλε χώρε. Με βάση όμω την μελέτη επιπτώσεων, που ήταν μια επίπονη προσπάθεια, έχω να σα πω, προέκυψε ότι αν τολμήσει η επιχείρηση να ξεμητήσει, πρέπει να πρέπει να δαπανίσει 70.153 ευρώ για να δραστηριοποιηθεί και στις 26 άλλες χώρες. Με αυτή την οδηγία τώρα, θα δαπανίσει απλώς 2.063 ευρώ. Κάτι παραπάνω από 2.000, Μία φορά θα δαπανίσει και τέρμα. Εμείς ως καταναλωτές τελικά πληρώνουμε την νύφη. Πρέπει να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες για να αυξήσουμε την ευημερία των καταναλωτών. Να μην οχυρωνόμαστε πίσω από προστατευτισμούς. Ο Ιρλανδός εκπρόσωπος ουσιαστικά μίλησε ανοιχτά για προστατευτισμό υπέρ των καταναλωτών. Έχετε υπόψη σας ότι όλες οι διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για προστατευτικούς σκοπούς. Όλες οι διατάξεις. Εάν δεν προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις βέβαια, με σωστό τρόπο, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Χρειαζόμαστε αυτή την ε, εσωτερική αγορά και τη χρειαζόμαστε να είναι σε καλή κατάσταση, σε εύρωστη κατάσταση. Πώς θα το καταφέρουμε χωρίς εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Πώς θα αισθάνθουν εμπιστοσύνη οι Ευρωπαίοι πολίτε ω καταναλωτέ σε άλλες χώρες. Αν δεν έχουμε κοινοτικά νομοθετήματα. Δώστε μου εσείς συμβουλέ. Βλέπω ότι αυτό το άρθρο 26 ε, που αφορά τις αποζημιώσεις και τις αποκαταστάσεις. Βλέπω ποια είναι η κατάσταση στην Ιρλανδία και, στην, και στον Αμήνο Βασίλειο. Μπορούμε να υπολογίσουμε. Αν επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση και αν οι καταναλωτές επιλέξουν το είδος της αποζημίωσης, εντάξει, θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή την ατραπό. Μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος της κάθε επιλογής, αν θέλετε. Αλλά οι διαφορές κοστίζουν. Και κάτι άλλο για τις εγγύησεις. Ο λιθωνός συνάδελφος ανέφερε το βάρος της απόδειξης. Ότι ο καταναλωτής έφερε αυτό το βάρος μέχρι τώρα. Και τώρα περνάει στον έμπορο. αυτή η προθεσμία είναι έξι μηνών. Το βασικό είναι η, το βάρος της απόδειξης να ισχύει για έξι μήνες σε ορισμένε χώρε έχουν μία προθεσμία 6 χρόνων προστασία και όχι 2 χρόνων. Το βασικό όμω είναι το εξάμεινο. Τώρα, αν ε, δεν σας αρέσουν αυτοί οι έξι μήνες, μπορούμε να του αυξήσουμε. Το θέμα δεν είναι ιδεολογικό. Μπορούμε να κάνουμε όποια επιλογή προτιμάτε. Το θέμα είναι τι κόστος θα έχει αυτό. Στις 15 Μαΐου θα πάμε στην Αυστρία. Ούτως ή άλλως επισκεφτώ όλα τα κοινοβουλιά σας. Θα είμαι σε επαφή μαζί σας. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ε, απαντήσεις που σας τις χρωστάω. Κυρία Καραμαλή από τη Γαλλία, σας ξέρω και προσωπικά, γνωρίζω τα διαφορετικά προβλήματα λόγω διαφορετικών ερμηνεών της οδηγίας. Είχα μια καλή συνάντηση με την Οργάνωση Προστασίας των Καταναλωτών στην Γαλλία πριν από 10 μέρες και συμφωνήσαμε ότι τα περισσότερα εκρεμή ερωτήματα αφορούν το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Και στην πραγματικότητα περί πρόκειται περί λανθασμένων ερμηνεών. Τους επόμενους μήνες θέλω να διευκρινιστούν κάποια θέματα. Δηλαδή η Γαλλία θα μπορέσει να κρατήσει το σύστημα που έχει για τους αθέμητους εμπορικούς όρους, για τα, τις κρυφές ζημίες. Μπορεί να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε τον κατάλογο. Ούτω ή άλλω μπορείτε να έρθετε σε Βρυξέλλες ε, και να τα συζητήσουμε αυτά για μισή μέρα. Να πω στο Σλοβαίνο συνάδελφο, στην κυρία από τη Σλοβενία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ θα έχουν το βέλτιστο δυνατό κοινό επίπεδο προστασίας για τις, τα μέσα αποκατάστασης ε, συνεχίζεται η συζήτηση, το είπα προηγουμένως, για τη συμπερίληψη των δημοσίων αρχών στον ορισμό του εμπορευόμενου. Το Συμβούλιο συζητάει αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα που το διαπραγματεύονται στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τμήμα της οδηγίας για τις εγγυήσεις για το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και το φυσικό αέριο που δεν ε, καλύπτονται από τις ε, διατάξεις για τις πωλήσει. Εδώ έχουμε κανόνες για τα άειλα αγαθά που δεν είναι κατάλληλε για αυτήν την περίπτωση. Αυτά τα συμβόλαια καλύπτονται από του κανόνες για τους αθέμητους ώρε, για την προσυμβατική ενημέρωση και ειδικού κανόνες για τι τις συμβάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και συμβάσεις που συνάπτονται εξ, Είναι μια αρχή, σα το είπα. Ελπίζω να είναι καλή αυτή η αρχή. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας για πρώτη φορά έχουμε ένα φόρουμ πολιτών που συζητάει τα θέματα ενέργειας και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τα τιμολόγια των προϊόντων ενέργειας και συζητάμε, κάνουμε συγκρίσεις τιμών για τις συμβάσεις ε, υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τη διάταξη για τις πωλήσει. Εδώ έχουμε κάποιες εξαιρέσεις οι εξαιρέσεις καλύψονται από τους κανόνες ε, για τους αθέμητους ε, όρους. Κύριε Τουμπον, η Κομισιόν πολύ σύντομα θα σας δώσει ένα πίνακα αναλύοντας κάθε θέμα, τις επιπτώσεις που έχει σε κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις επιπτώσεις ε, της οδηγίας στους εθνικούς κανόνες και στην εθνική νομοθεσία. πολλά προβλήματα θα εξανεμιστούν, πολλοί μύθοι θα καταπέσουν και κάποια πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Κυρία Ριπέλοβα, για το CFR, η πρόταση είναι αποτέλεσμα μακράς διαδικασίας διαβούλευσης και το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα συνεχίσει να είναι πηγή έμπνευση. Το πλαίσιο αυτό είναι ουσιαστικά μια εργαλειοθήκη για την ε, αναθεώρηση του κεκτημένου για τους καταναλωτές. Ε, είχαμε πολλά εργαστήρια ε, και σε πολλούς τομείς το πλαίσιο αναφοράς ουσιαστικά λειτουργεί. Παράδειγμα Παραδείγματο χάρη, το πλαίσιο αυτό μα οδήγησε στο να εισαγάγουμε τον λεγόμενο μαυροπίνακα για του αθέμητου όρου και τι αθέμητε πρακτικέ. δεν σε ικανοποιεί όλου, αλλά είναι CFR ο ορισμός ε, της ε, μεταφοράς του κινδύνου, προσυμβατικής ενημέρωσης κτλ. Οι Σλοβαίνοι, οι Έλληνες, οι Σουηδοί συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει επίπεδο προστασίας υψηλό και πιο φιλικό για τους επιχειρηματίες. Έτσι πρέπει να συμβαίνει. Αποκλείεται να κινηθούμε Μειώνοντα την προστασία του καταναλωτή. Θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά την προστασία ε, για να υπάρχει συνένεση και εμπιστοσύνη των καταναλωτών χωρίς να επιβάλλουμε παράλογα, παράλογες δαπάνες σε επιχειρήσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα των εγγυήσεων και της αποκατάστασης, της μεταφοράς του κινδύνου και πώς μπορούμε και εκεί να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας. Κυρία Πιστρέλο. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρότασή σας. Θα συζητήσουμε πολύ σύντομα όταν έρθω στη Ρώμη. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, γιατί χρειαζόμαστε και ενθάρρυνση στην ομάδα μου. Ο κύριος από την Πολωνία. Ζητώ συγγνώμη που τα προφέρω λάθος τα ονόματα. Συμφωνώ μαζί σας ότι Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να μην βαρύνουμε υπερβολικά τι επιχειρήσει και να προστατεύσουμε παράλληλα και του καταναλωτέ Για τη διαβούλευση με του καταναλωτέ. Οι υπηρεσίε μου και εγώ είχαμε ευρείε διαβουλεύσει με τους οργανώσει των καταναλωτών ε, και είχαμε κυκλοφορήσει μια πράσινη βίβλο πριν αναθεωρήσουμε την οδηγία. Επομένω η βίβλο αυτή έχει κυκλοφορήσει. Ε, είχαμε 400 απαντήσεις στην πράσινη βίβλο προς τους αυστριακούς συναδέλφους. Με βάση την ε, επισκόπηση που κάναμε, το 70% των εμπόρων δεν πουλάνε διασυνοριακά γιατί δεν υπάρχουν αρμονισμένοι κανόνες. Ε, αν υπάρχει πραγματική ενιαία αγορά, θα υπάρχει ε, καλύτερη, μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές, φθηνότερες τιμές κτλ δεν θα κάνω κανένα συμβιβασμό στη δημιουργία μιας αγοράς για τους πολίτες. Και θέλω πραγματικά να υπάρχει μία δέσμη κανόνων και για τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αφήσω κόπον για να κάνω ό,τι μπορώ στα πλαίσια αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ για αυτή την υποστήριξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για μια αγορά για τους καταναλωτές. Είμαστε στη δεύτερη φάση ολοκλήρωσης της ενίας αγοράς. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνα των καταναλωτών, γιατί οι καταναλωτές διαμορφώνουν την οικονομία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κάνουν στο παρελθόν. Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω να κάνω το καταδύναμη και πάνω από αυτό. Πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε θα τα καταφέρουμε. <laughs> Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούνεβα για τις απαντήσεις σας. Πολλές ερωτήσεις. Εκτιμώ πολύ ότι εμβαθύνατε και στις απαντήσεις σας, λεπτομεριακά απαντήσετε και καλό θα ήταν να στείλουμε όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι μόνο στις αρμόδιες επιτροπές. Θα ήθελα να ε, δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο και φίλο από την Τσεχική Γερουσία για να ολοκληρώσει ένα σύντομο τελικό σχόλιο. Uh, uh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση και πολύ γόνιμη. Μάθαμε ε, τα πρόσφατα σχέδια των διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί πολλή χρόνο για τις διαπραγματεύσεις και εύχομαι ε, κάθε επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα κληθεί να αξιολογήσει και να συζητήσει διάφορες αποκλίνουσες απόψεις. Ακούσαμε πως έχει κατάσταση των πραγμάτων σε διάφορα κράτη-μέλη πολύ χρήσιμο είναι αυτό για τους καταναλωτές διότι αυτό που χρειάζεται είναι νομική ασφάλεια. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες. Μήπως χαλαρώσει η προστασία των καταναλωτών εκεί που είναι πολύ υψηλή. Μήπως αποδυναμωθεί. Τι γίνεται με την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που ε, θίγονται. Αυτά είναι ακόμα ε, ενδεχομένω κάποιε ελλείψεις στην οδηγία, κάποια παραθυράκια που πρέπει να κλείσουν. Ορισμένοι συναδελφοί αναφέρθηκαν στην αρχή τη επικουρικότητα. Ακούσαμε επίση ότι χρειάζεται ε, μια ενιαία εναρμόνιση ε, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βρούμε και τη σωστή ισορροπία από τη μια να προστατεύουμε τους καταναλωτές και από την άλλη να ε, προστατεύουμε τις επιχειρήσεις. Βλέπω ότι η Επίτροπός μας ε, ε, έχει πολύ ενθουσιασμό και ελπίζω να πετύχει. Και σας εύχομαι σε όλους καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Τόνισε ο συνάδελφος πως το σημαντικότερο για μας είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Πράγματι. Και αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Παρακαλώ 3 και 40, 3 και μισή μάλλον. Παρακαλώ να είστε πίσω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Έξω έχει καφέ. Uh,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 AUTHORWAVE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 Who dear we need to start. please take your seats. Συνάδελφοι, thank you very much that you will, you will... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιστρέψατε και για τη δεύτερη συνάντηση, της διακοινοβουλευτική μας συνάντηση. Θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω τον, τη συνάδελφό μου Σόνια Παρκούτοβα από την Τσεχική Γερουσία να μας καλωσορίσει. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας μετα δώσω τους χαιρετισμού της ε, τσεχικής γερουσίας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και δεν νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη που θα πει ότι αυτή η διακοινοβουλευτική συνάντηση που διοργανώνονται από την Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι κάτι το πολύ θετικό, γιατί είναι σημαντικό να συζητηθεί η οδηγία και ανυπομονώ να ακούσω και τις ε, υπόλοιπες συζητήσεις μας. Ναι, λέει η Πρόεδρος, ο χρόνος ε, τρέχει, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Orwells από την νομική σχολή του Μάντσεστερ που ειδικεύεται στο δίκαιο των καταναλωτών. Θα ήθελα να μας ε, παρουσιάσετε τα σχόλιά σας, τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας για την εφαρμογή και το μέλλον του Τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών στην εθνική νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Μετά την παρουσίασή σα. θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσει. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ο It's είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ ως μη πολιτικός για να μιλήσω σήμερα, αλλά αυτό αποτελεί και μία ευθύνη το γεγονός ότι είμαι ο μόνος μη πολιτικός και είναι πολύ δύσκολο κατά κάποιο τρόπο να συζητήσουμε θέματα εφαρμογής ε, μεταφοράς ε, του, της νομοθεσίας αυτής για σε 20 λεπτά μόνο. Θα παραλείψω κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες μπορείτε να θέλετε να διευκρινίσω. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές που προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά, αλλά ήθελα να δώσω και κάποια παραδείγματα για τις ε, τέσσερις ε, οδηγίες που καλύπτονται από ακούσαμε και σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις σε αυτό το πρόβλημα. Τα θέματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό και σε ό,τι αφορά την εγχώρια εφαρμογή του κεκτημένου αυτού και η τρίτη πτυχή είναι η σχέση μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης εναρμόνισης. Και κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, θεωρητικά είναι το πιο ενδιαφέρον και δύσκολο αυτό το τελευταίο στοιχείο. Γιατί πολλά στοιχεία από αυτά που βλέπουμε στο κοινοτικό κεκτημένο μπορούν να τροποποιηθούν κάνοντας ε, τα πράγματα καλύτερα στο μέλλον αλλά η επιλογή μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης συναρμόνισης είναι πραγματικά κάτι το θεμελιώδες για τη σχέση μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Και επίση κάτι το οποίο ίσως γίνεται λιγότερο κατανοητό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό καθορίζει και τις σχέση σε εταιρικό επίπεδο μεταξύ του δικαίου του καταναλωτών και του γενικού συμβατικού δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση. Να εξηγήσω λοιπόν καταρχά κάποια από αυτά τα θέματα για το ευρωπαϊκό κεκτομένο, την εσωτερική εφαρμογή και μετά να εστιαστούμε τη συζήτησή μα για την μέγιστη εναρμόνιση. Ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ανάγκη να υπάρξουν κάποιοι ορισμοί κοινοί σε όλες αυτές τις οδηγίες. Στις τέσσερις συγκεκριμένες οδηγίες, δηλαδή, που θα πρέπει να εναρμονιστούν με την παρούσα πρόταση. Απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα τι είναι η ημέρα, η περίοδος απόσυρσης. Πράγματα που νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι καλά θα κάνουμε να τα εναρμονίσουμε και αν εναρμονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πιο πολλέ οι πιθανότητε ότι θα διαμορφωθεί με παρόμοιο τρόπο και το εθνικό δίκαιο, γιατί σε εθνικό επίπεδο έχουμε τον πειρασμό να διορθώνουμε πράγματα τα οποία είναι σφαλμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό νομίζω ότι θα λύσει και διάφορα κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τα οποία επί του παρόντο καλύπτονται δηλαδή από το εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει να πω ότι πολλά από τα παραδείγματα που έχω τα βρήκα σε ένα παράρτημα το οποίο δημοσιεύτηκε βάσει έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, σας συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό το με αυτό το παράρτημα, το οποίο παρουσιάζει λεπτομερώς ε, ποιες είναι, είναι τα κενά στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, να σας μιλήσω και για τη χρήση των γενικών ρητρών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Καταρχάς, επειδή και το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να πω ότι οι γενικές ρήτρες αποτελούν νέο φαινόμενο για μας. Είχαμε μία απόφαση που όριζε, για παράδειγμα, την καλή πίστη, που θα μπορούσε να δεχτεί κριτική, ότι δεν κατανοούμε δηλαδή σωστά την, ε, τον όρο αυτό. Ωστόσο υπάρχει και ο εξίσου μεγάλος ε, κίνδυνος αν υπάρχει ερμηνεία σε εθνικό επίπεδο για του όρου αυτού, να του ερμηνεύουμε έτσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι διαπιστώνουμε ότι 7 κράτη-μέλη δεν συμπεριέλαβαν την καλή πίστη στα εθνικά του σχέδια. Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο προβληματίστηκε Δηλαδή πώ θα χρησιμοποιήσουμε έναν όρο ο οποίο δεν χρησιμοποιείται σε 7 από τους εφαρμοστικού νόμου. Και σε κάποιο βαθμό να σα ρωτήσω και το εξή Μπορεί να γίνει εναρμόνιση βάση γενικών ρητρών. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Hofstadt είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αυτό που λέει είναι ότι η κατανόηση του κατά πόσο ο σκοπός είναι αθέμητος θα πρέπει να γίνεται σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου και του εθνικού νομικού περιβάλλοντος, το οποίο συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφορικά με το συμβατικό δίκαιο που επηρέασε και τη θεμητότητα του σκοπού. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η εναρμόνιση βάσει της γενικής αυτής ρήτρας θα έχει πρακτικά αποτελέσματα και ωφέλειες Όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για παράδειγμα θα κοστίσει λιγότερο η όλη διαδικασία, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται ίσως για απλούστευση του προβλήματος. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ασφαλώς, υπάρχουν ασφαλώς πολλές διαφορετικές ρυθμιστικές παραδόσεις. Κάποιες ε, χώρες προτιμούν το αστικό δίκαιο, κάποιες άλλες το ποινικό, κάποιες το δίκαιο αυτορύθμισης και προφανώς πρόκειται για μέρη του, της γενικότερης νομοθεσίας, αλλά έχουμε εθνικές νομοθεσίες για το πώς εφαρμόζεται το δίκαιο και υπάρχουν και αποφάσεις του ΔΕΚ φυσικά, που λένε για παράδειγμα ότι η Ολλανδία δεν ε, εφήρμοσε στο αστικό του δίκαιο ανάλογα το υφιστάμενο δίκαιο και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές παραδόσεις για το οποίο θα συνεχιστεί και στο μέλλον κατά πάσα πιθανότητα. We've got examples of blatantly incorrect implementation. Και φυσικά έχουμε και πολλά παραδείγματα απλά εσφαλμένης εφαρμογής ή διαφορετικής ερμηνείας του τι ζητά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή αυτό δια, φυσικά διαφέρει από κράτο σε κράτο και από οδηγία σε οδηγία. Ωστόσο, θα θέλαμε να πω ότι κάποιε φορέ η καθυστέρηση αυτή αποτελεί απόρρια της προσπάθειας να γίνει καλή δουλειά στην εφαρμογή του νόμου. Και αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε σε ό,τι αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, στην, στον Εμένο Βασίλειο, που είναι μεγάλη δουλειά αλλά διήρκησε πάρα πολύ χρόνο. I'm a little bit concerned about in some of the language I've heard in the documentation I've read. Κάτι άλλο που με είναι η κριτική του εθνικού δικαίου ότι χρυσώνει το χάπι. γιατί μπορεί κάποιοι να λένε ότι υπερβάλλει το εθνικό δίκαιο, αλλά κάποιοι ακαδημαϊκοί θα μπορούσαν να πούν ότι προσπαθεί απλά το εθνικό δίκαιο να βρει τον καλύτερο τρόπο εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκούμε. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία για τον αντίκτυπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Το επίπεδο προστασία των καταναλωτών σε πολλά κράτη, σχεδόν σε κάθε κράτο, είναι πολύ καλύτερο σήμερα, ακριβώ λόγω του αντίκτυπου τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και πολλέ από τι θεμελιώδει ελευθερίε μα έχουν εναρμονιστεί. Υπάρχουν φυσικά λεπτομέρειε οι οποίε ακόμα διαφέρουν, αλλά γενικέ γραμμέ έχουν εναρμονιστεί. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές κοινείς ε, αντιλήψεις ε, στην προστασία των καταναλωτών και θα μπορούσαμε όντως να πουλήσουμε, αν θέλετε, αυτό το μοντέλο ως ένα συνολικό πακέτο. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και των εθνικών αρμοδιοτήτων. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι κατά πόσο θα κοιτάξουμε μόνο την προστασία των καταναλωτών, το συμβατικό δίκαιο ή μήπως θα έπρεπε να υπάρξει μια γενικότερη εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών δικαίων, δηλαδή να ενταχθεί στο και το αστικό και το ποινικό δίκαιο στα πλαίσια του συμβατικού δικαίου. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν αν είναι σημαντικό αυτό για μας, αν θεωρούμε δηλαδή ότι το δίκαιο για τους καταναλωτές θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο. Τώρα να σας παρουσιάσω την πρώτη μου περίπτωση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας αθέμητων πρακτικών. Βλέπουμε εδώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο για το πώς αντιμετωπίζουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. 22 νόμους ε, τροποποιήσαμε για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ακόμα και νομοθεσίες του 1968 καταργήθηκαν και εισήγαμε τις γενικές ρήτρες. Γενικά νομίζω ότι ήταν θετική η εφαρμογή της οδηγίας και ήταν και καλή η αποδοχή, αλλά εξακολουθούν να επικρατούν κάποιες αμφιβολίες για θέματα ερμηνείας της οδηγίας και σε ό,τι αφορά τις γενικές ε, ρήτρες και τις επιθετικές πρακτικές και του καθεξής. Διάβασα τον προηγούμενο μήνα μία παρουσίαση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί σημειώθηκε μείωση των ενστάσεων από τις τοπικές υπηρεσίες και είπαν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Άρα, ίσως να είναι λιγότερο εύκολο πλέον για τις υπηρεσίες αυτές να εφαρμόσουν στην πράξη τη νέα νομοθεσία. Άρα θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο πρακτικός αντίκτυπος της πρότασης, αν θα είναι επωφελής, αν είναι θετικός ο αντίκτυπος. Η οδηγία για τις αθέμητες ε, εμπορικέ πρακτικές και για την παραπλάνηση είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργείται μια οδηγία μέγιστης εναρμόνισης για την προστασία των καταναλωτών. Αλλά στο business to business, επίπεδο επιχειρήσεων προεπιχειρήσεων, έχουμε ελάχιστη εναρμόνιση. Δηλαδή, οι καταναλωτέ χρειάζονται το μέγιστο επίπεδο εναρμόνιση και οι επιχειρήσει όχι. Χρειαζόμαστε κάποια εξήγηση εδώ. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό απομονώνει, αν θέλετε κάπως, το δίκαιο για την προστασία του καταναλωτή. Θέλουμε δηλαδή τι, να το διαχωρίσουμε από το υπόλοιπο δίκαιο. και υπάρχει μια πολύ καλή σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση που καταδεικνύει διάφορες προσεγγίσεις για την εφαρμογή σε κάποιες χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία όπου υπήρχε παλιά μία ισχυρή γενική ρήτρα που καλύπτει και τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών μάλλον επιχειρήσεων καταναλωτών και επιχειρήσεων επιχειρήσεων, διατηρήθηκε και στο εθνικό δίκαιο αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση, το οποίο σημαίνει ότι το εθνικό δίκαιο φυσικά δεν εναρμονιζόταν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο κάνει αυτή τη διάκριση μεταξύ business to business και ε, business to consumer. Άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία, αναφέρω παραδείγματα, εφήρμοσαν συγκεκριμένα τους νόμους για τους καταναλωτές. Και εκεί προκύπτει αυτή η απομόνωση, αν θέλετε, του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αναφέρω σε λίγο. Say that the European Commission Νομίζω πως αληθεύει αν πει κανεί ότι η Κομισιόν ήταν πολύ ικανοποιημένη με την οδηγία για τις δίκαιες εμπορικές πρακτικές, το πώς κατάφεραν την εναρμόνιση και θέλουν αυτό να το ξανακάνουν στο πλαίσιο της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Βλέπουν προβλήματα κατάλληλη εφαρμογή. τα κράτη-μέλη ε, πολλές φορές ε, περιορίζουν το πεδίο εφαρμογή στην εφαρμογή των μέτρων και παίρνουν, ε, κάνουν κάποιες επιλογές και χρησιμοποιούν την ρήτρα ελάχιστης εναρμόνισης. Και όλα αυτά τα παράδειγματα που δίνω ε, έχουν ε, αναφερθεί στο κομπέντιουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ε, δίκαιο του καταναλωτή. Να σας πω λοιπόν καταρχήν τι συμβαίνει αν τα κράτη-μέλη ξεπεράσουν το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα. Επιτρέπεται να το κάνουν. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με το πλαίσιο. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Ας πούμε ότι η οδηγία τελικά καλύπτει μόνο προδιατυπωμένα στάνταρ, προδιατυπωμένες συμβάσεις. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν τους δικούς τους ελέγχους στα, ε, στις συμβάσεις ε, τις ατομικές. Ε, εδώ τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να τα ξεπεράσουν. Αν όμως πάρουμε την οδηγία ε, για τις κατοίκων πωλήσει που συμπεριλαμβάνει πωλήσει λιγότερο των, ε, χαμηλότερα των 60 ευρώ, μπορούν τα κράτη-μέλη να το ξεπεράσουν αυτό και να πάνε κάτω από τα 60 ευρώ. Εγώ νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν προβληματικό, διότι το εμπόριο μπορείς να το ε, ελέγξεις, να το ρυθμίσεις μέχρι τα 60 ευρώ, αλλά ίσως ένα κρατομέρες μέλος να επιλέξει να κατεβεί κάτω από τα 60 ευρώ. Αυτό επιτρέπεται, η Κομισιόν το κάνει, το επιτρέπει, η οδηγία είναι δεσμευτική για τα κρατημέλη όταν μιλάει για πωλήσει μέχρι 60 ευρώ. Και τελικά το παράδειγμα που είχαμε σήμερα το πρωί, η ιδέα ότι από τη στιγμή που έχουμε την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, αυτό μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το, την ε, γνήσια σύμβαση με βάση την νομοθεσία οι Γάλλοι, ίσως μπορεί να είναι ευχαριστημένοι αν διατηρήσουν το βίσκασε, αλλά πώς είναι αυτό συμβατό με την οδηγία για την μέγιστη εναρμόνιση. Εγώ δεν είμαι υπέρ της maximum εναρμόνισης, αλλά δεν νομίζω πώς μπορούμε, ότι μπορούμε να λέμε ε, ότι σκοπεύουμε στην μέγιστη εναρμόνιση, ενώ επιτρέπουμε την χρήση του, της εθνικής νομοθεσίας. Έχουμε κράτη-μέλη και ανησυχεί, ανησυχεί για αυτό ότι τα κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει την ελάχιστη δυνατή εναρμόνιση και θέλουν να δημιουργήσουν μια πιο ομοιόμορφη, εναρμονισμένη εθνική, μάλλον ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπορεί αυτό να γίνει. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποιες πτυχές όπου μπορεί να γίνει. Μπορεί δηλαδή κανείς να δημιουργήσει ομοιόμορφη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ίσως ε, να μπει σε, κάποιες, ε, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς όπως ας πούμε η ενημέρωση ή τα δικαιώματα απόσυρσης, μπορεί όλα αυτά να μπορούν να εναρμονιστούν με τυποποιημένο τρόπο. Όμως, όποιο μεγαλύτερη σύνδεση έχει ε, μια, ένας τομέας του δικαίου με το εθνικό δίκαιο είναι τόσο πιο δύσκολο να διατηρηθεί η, ο έλεγχος, ε, τόσο πιο δύσκολο να ελεγχθεί η εφαρμογή του συμβατικού δικαίου. Και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου οι καταναλωτές μπορεί να μην θέλουν να τους μεταχειρίζονται ως καταναλωτές στο δικό τους νομικό σύστημα. Εγώ έχω προσπαθήσει να μην δώσω εθνικά παραδείγματα εκτός από τη δική μου χώρα, γιατί δεν θέλω να μπω ε, στα χωράφια άλλων ειδικών στην αίθουσα και είμαι βέβαιος πως η πολωνική αντιπροσωπεία θα με διορθώσει αν δεν κατάλαβα καλά την Πολωνία. Αλλά σας δώσω ένα παράδειγμα σε μια πρόσφατη διάσκεψη που διοργανώθηκε και ένα παράδειγμα που έδωσε ο καθηγητής Ζόργ. Ε, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο έχει ε, εκείνος εκδώσει και αυτό που μας είπε είναι ότι όταν η Πολωνία επέλεξε να εφαρμόσει την οδηγία για τις πωλήσει, το έκανε μέσω ενός ε, μεμονωμένου συνόλου κανόνων και συνέπεια ήταν ότι συχνά ένας καταναλωτής είναι σε καλύτερη θέση όταν βασίζεται στην ε, πολωνική νομοθεσία παρά στην ε, οδηγία. Και το ερώτημα ήταν, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να αρνηθούν το καθεστώς τους ως καταναλωτές. Τέτοιες ερωτήσεις δυστυχώς ε, δεν επιτρέπονται γιατί οι καταναλωτές, γιατί θεωρείται ότι προσπαθούμε να αφαιρέσουμε δικαιώματα. Αλλά οι καταναλωτέ, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, μπορούν να αρνηθούν αυτό το καθεστώ. Αυτή ίσως να είναι μια λύση που μπορεί να την έχουν οι καταναλωτέ αν η οδηγία εφαρμοστεί με ε, τη σημερινή της μορφή. Αν πάρουμε το δικό μου, τη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα, όπου έχουμε εγώ έχω δύο ανησυχίες για τις διατάξεις για τις πωλήσει που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Καταρχήν ότι χάνουμε το αυτόματο δικαίωμά μας για να απορρίψουμε κάποιο αγαθός και έπειτα έχουμε ένα νέο καθήκον να ενημερώσουμε τον πολιτή μέσα σε δύο μήνες από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αυτό δεν θα εφαρμοζόταν αν είχα τη γενική νομοθεσία για τις πωλήσει, αλλά θα ίσχυε αν έπρεπε να εφαρμόσω την οδηγία. Μπορώ να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να θεωρούμε καταναλωτής και να θεωρούμε ως επιχείρηση αν αυτό συμβεί σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα είναι καθόλου καλό για την προώθηση και τη ε, ε, διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προστατή των ε, καταναλωτικών δικαιωμάτων, αν οι καταναλωτέ θέλουν να επιλέξουν ότι θα μείνουν εκτός του καθεστώτος του καταναλωτή, του ευρωπαϊκού καθεστώτος του καταναλωτή και ότι θα επιλέξουν το καθεστώ για τι επιχειρήσει. Για αυτό το θέμα της εναρμόνισης πιστεύω πραγματικά πως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή πολύ περισσότερο στο διαφορετικό πλαίσιο εντός του οποίου γίνονται τα διάφορα επιχειρήματα. Υπάρχουν κάποια πλαίσια όπου συμφωνώ απολύτως ότι η μέγιστη εναρμόνιση θα είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, ε, για τους κανόνες και τη σύσταση των προϊόντων, η ετικετοθεσία, διαφήμιση, ακόμα και τυποποιημένες συμβάσεις, ε, όπου μάλλον μάλλον χρειάζεται ο κανόνας της μέγιστης εναρμόνιση. Ορισμένοι δηλαδή συμφωνούν ότι θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή μαύρη λίστα. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι κανόνε που πρέπει να εναρμονιστούν, όπω το δικαίωμα απόσυρση ή το καθήκον για ενημέρωση, πληροφόρηση. Όμως αυτό αυξάνει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης πληροφόρησης υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα στην οδηγία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου η οδηγία έπρεπε να συμπεριλάβει 32 υποχρεώσεις πληροφόρησης που συλλέχθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτοί οι γενικοί κανόνες δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα του, της, αγοράς σε μια χώρα, απλώς ε, περιθωριακά επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που δεν χρειάζεται να εναρμονιστούν. What Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα εδώ όσον αφορά την μέγιστη εναρμόνιση. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και υπάρχει και σοβαρό κόστο και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πω αξίζει να πληρώσουμε αυτό το τίμημα. Και γι' αυτό και με ενθαρρύνει αυτή η συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, όπου είπαμε ότι μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάποιε υποχωρήσει από τη στιγμή που είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει ένα πραγματικό απτή βελτίωση στην εσωτερική αγορά που γενικά θα ωφελήσει τους καταναλωτές. θα έχουμε μία ε, γενική προστασία για τους καταναλωτές που μπορεί να είναι χαμηλότερη και η νομοθεσία για τον καταναλωτή θα περιοριστεί στην ευρωπαϊκό αυτοκαθεστώς. Το ρίσκο της υπερβολικής ε, ε, ρύθμισης υπάρχει ως αποτέλεσμα όλων αυτών των συμβασμών και πραγματικά υπάρχει και κίνδυνος ότι μπορεί οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν προβλήματα στα οποία δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε αρκετά γρήγορα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία. Πολύ σύντομα για την επιβολή της νομοθεσίας, Πρόεδρε, πέντε λεπτά και ακόμα. Όταν μιλάμε για την ε, πραγματική επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή πόσο μπορούμε να είμαστε σοβαροί για μια πλήρη ομοιομορφία νομοθεσίας όταν βασίζουμε πολλές από αυτές τις αρχές σε γενικές, αρχές, σε γενικές ρήτρες που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο των διαφορετικών παραδόσεων στην Ευρώπη, διαφορετικέ δυνατότητε πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ακούσαμε χθε πώ στη Γερμανία είναι δυνατόν να μέσα σε μια μέρα να κάνει κανεί την καταγγελία για παραπλανητική διαφήμιση, αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκο από υπό άλλα υπό άλλα εθνικές νομοθεσίες. Αυτή τη στιγμή είναι μια καθολική τεχνική ε, που χρησιμοποιείται κατά της παραπλανητικής διαφήμισης. Αλλά πώς εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπηρεσία για το δίκαιο εμπόριο ε, προσπαθεί να κάνει κάτι για τις ε, παραπλανητικές συμβάσεις και θέλει να προβεί σε κάποιους αφαιρημένους ελέγχους που λέει ότι ναι, οι όροι επιβεβαιώνονται αόριστα, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά οποιοδήποτε υπάρχοντος ε, καταναλωτή. Και η απάντηση του Ανώτου δικαστηρίου ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για μεμονωμένες συμβάσεις, γιατί πάντοτε μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τη χρήση Ενό ενός όρου που μπορεί αντικειμενικά να είναι άδικος. Αν εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον στον Ηνωμένο Βασίλειο πολύ λίγο νόημα θα έχει το να έχουμε έναν αφηρημένο έλεγχο των άδικων όρων. Γιατί το νόημα του αφηρημένου ελέγχου τι είναι ότι μπορείς να... Ποιο θα είναι από τη στιγμή που μπορείς να, να, να υποστηρίξεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο όρο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Άλλες χώρες μπορούν να ακολουθήσουν άλλη πορεία. Πολύ διαφορετικές ε, προσεγγίσεις δηλαδή στην πρακτική εφαρμογή της... Ε, ε, άμεσων διαταγών. ή των δικαστικών εντολών. Επίσης, η των δικαστικων εντολων Επίση, η σημασια του αστικού δικαίου σε αντίθεση με το ποινικό. Σε ορισμένε χώρες οι αθέμητε εμπορικές πρακτικές δίνουν ε, λαβή για απαιτήσει αποζημίωση. Στον Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται. Δεν ε, μπορεί να κάνει κανείς ενέργειες για τις αποζημιώσεις. Εκεί βασιζόμαστε στο ποινικό δίκαιο ή σε δικαστικέ εντολές. Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστούν οι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, ώστε να έχουν μια πιο ευρωπαϊκή προοπτική. Να βρούμε δηλαδή έναν τρόπο με τον οποίο το διασυνοριακό πρόβλημα να, να ξεπερνά την εθνική ατζέντα. τμήμα του προβλήματος είναι το να ελέγξουμε τα διάφορα επίπεδα προστασίας. Γιατί αυτό που το οποίο εγώ είναι ότι σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου έχουμε ε, γραφεία ελέγχου σε κάθε πόλη, η συνεργασία ανάμεσα στην εθνική κυβέρνηση και στις Βρυξέλλες φαίνεται πολύ απομακρυσμένη. Πώς λοιπόν βλέπουμε την σημασία όλων αυτών όταν έχουμε να κάνουμε με τοπικά θέματα, θέματα της πόλεις μας, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προβλήματα αυτά προωθούνται προς τις εθνικές κυβερνήσεις και μετά στις Βρυξέλλες. Πώς δηλαδή θα εμπλακούν όλοι αυτοί. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε θέματα ε, συνεργασίας μπορεί να πρέπει να αγκαλιάσουμε τον κόσμο που επιτόπου δουλεύει για την επιβολή της νομοθεσίας, που μπορεί να μην είναι τελικά τα εθνικά ε, σώματα. Θα ήταν ευκολότερο ίσως αν υπήρχε κεντρικό σύστημα επιβολής νομοθεσίας. Και γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ε, αφού αυτό δεν υπάρχει, μια ευρύτερη προσέγγιση. Νομίζω πως έχω ξεπεράσει το χρόνο μου και εγώ θα ήθελα να ακούσω τις εθνικές προοπτικές και την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε για την Βρετανική νομοθεσία, το Βρετανικό δίκαιο. Εγώ Θα ήθελα να κάνω διάφορα σχόλια από την άποψη μιας πρώην γερουσιαστού για τα νέα κράτη-μέλη που δεν είμαστε τόσο νέα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πριν από έξι χρόνια εναρμονίσαμε πολύ γρήγορα την νομοθεσία μας και θυμάμαι πως για παράδειγμα οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ήταν πολύ σημαντικές όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν υιοθετήσαμε αυτή την, εδώ την οδηγία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, την υιοθετήσαμε στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρεπόταν από την Κομισιόν. Και πιθανότατα το ίδιο συνέβη και για άλλα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το μισό της ε, Ένωσης έχει εναρμονίσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα θέματα καταναλωτή από ότι τα παλιότερα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και για μας είναι πολύ σημαντικό το να βρεθεί μια σωστή ισορροπία ώστε να εναρμονιστεί η νομοθεσία για τον καταναλωτή και να είναι κατανοητή για όλους στην Ένωση. Διότι η διασυνοριακή αγορά είναι ακριβώς ένα από τα πλεονεκτήματα της Ένωσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω για την μεταφορά της οδηγίας ο συνάδελφος να μας κάνει κάποια σχόλια από την Επιτροπή Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να παραδεχθώ ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στα οποία έχω συμμετάσχει εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια είναι η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Θα αρχίσω με ένα γενικό σχόλιο και συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως. Και προηγουμένω συζήτηση φαντάζομαι, δυστυχώ δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Παρακαλώ να συμπληρώσετε τα έντυπα που σας ε, έχουν διανεμηθεί για να ξέρω ποιοι θέλουν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αγορητών. Νομίζω ότι θα πρέπει το, Εθνικό, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια να ασχοληθεί περισσότερο από... με την ε, οδηγίες αυτές καθώς και με την ερμηνεία τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια εμπειρία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλους και ίσως έγινε κάπως ενωρίς. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας εσείς. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε με όλες τις πληροφορίες που είχαμε και τα αυτό το οποίο κάναμε, εάν πραγματικά μετά από αξιολόγηση που έγινε υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε. θα κάνω κάποιε παρατηρήσει για να πιω ποια είναι η προσθέμενη αξία και θέλω να ακούσω και του συναδέλφου από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα. Αυτό που προσπάθησε να κάνει για το SWIP η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή για το Airline sweep και το Ringtone sweep όπως αναφέρονται πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με το στοιχείο το διασυνοριακό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως διότι το δίκτυο προστασίας των καταναλωτών διασυνορικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η πρακτική διαφέρει ένα κράτο και όντως πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να εξετάσουμε αυτό το θέμα πιο προσεκτικά, δεδομένου ότι δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά τα νέα κρατημέλη βεβαίω χρειάζονται περισσότερη συνδρομή για τέτοιου θέματα. Σωστά είπε η κυρία Ρόιτοβα ότι στην ε, διαδικασία διαπραγματεύσεων οι χώρες μας έπρεπε να χειριστούν ε, ε, βουνά νομοθεσίας για τα διάφορα θέματα και όντως υπάρχουν και να ε, υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ε, κανονισμών και οδηγιών κοινωτική νομοθεσία γενικότερα στην οποία πρέπει να συμμορφωθούμε. Κάτι άλλο το οποίο πιστεύω ότι επίσης είναι σημαντικό σε αυτήν την έκθεση είναι ότι αναφέρει κάτι το οποίο θέλει να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δίκτυο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθεί, είναι απαραίτητο για να γνωρίζουν οι πάντε πώ έχουν οι εμπορικές πρακτικές και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε. Και τελευταίο, όχι λιγότερο σημαντικό, νομίζω ότι ίσω έχουμε μία χρονική καθυστέρηση στο ότι θα πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές για τα δικαιώματα τα οποία έχουν. Πολύ συχνά μιλούμε για εκστρατείες ενημέρωσης, λέμε πάντα τι θα πρέπει να κάνει η Κομισιό, τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι κυρίως τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη όχι μόνο να ενημερώσουν, αλλά δώσουν και κάποιες γενικές οδηγίες στις επιχειρήσεις του σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης, αντιστοίχως, η Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βελτιώσει το θέμα αυτό. Να δημοσιεύσει μικρούς οδηγούς ε, για να ενημερωθούν καλύτερα και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. αναφέρθηκε κάτι το οποίο κάνει η Αγγλία και πιστεύω ότι είναι ίσως ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι για θέματα ενημέρωση. Επίσης, εξετάζοντας την ε, μεταφορά, την εφαρμογή και θέση σε εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών σε εθνικό δίκαιο θα πρέπει να δούμε είναι η κατάλληλη στιγμή έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε μια checklist και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινοβουλίων, για να βοηθηθούμε εξετάζοντας όλα αυτά τα θέματα, διότι όταν πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση για να δούμε πώς εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο και σε όλη την Ευρωπα... του καθενός και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να γνωρίζει το θέμα πολύ καλά και θα πρέπει να έχουμε όλη την ίδια μέθοδο αξιολόγηση, τα ίδια εργαλεία για να δούμε εάν εφαρμόζεται η κάθε κοινοτική οδηγία κανονισμό στο εθνικό δίκαιο. Γιατί για να κάνουμε συγκριτικές αναλύσεις πρέπει να ακολουθήσουμε παρεμφερείς διαδικασίες και μέσα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I would like to ask... Uh, Θα ήθελα να, ευχαριστήσω, ε, ευχαριστήσω και να ζητήσω τώρα από μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων να μας μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία όσον αφορά γενικά την μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό σας δίκαιο. Και επίσης παρακαλώ συμπληρώστε το σχετικό χαρτί για να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο αγοριτών. Η συμπρόεδρος επίσης θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Τι αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέγονται για την μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στα εθνικά δίκαια αναφέρονται οι γενικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε και βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα που είναι συζητήσιμα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ποια είναι η θέση των διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση με το πώς έχει η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Πρέπει να πω τουλάχιστον στη δική μα περίπτωση στη χώρα μα είναι κάπω παθητική η στάση τη δική μα βουλή, Διότι η κυβέρνηση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μεταφορά και η εφαρμογή τη οδηγία, του νέου νόμου, τι νέε νομοθετικέ πράξει για να γίνει η μεταφορά τη κοινότική οδηγία. Η Κατοβουλή και η Γερουσία στην Τσεχία εξετάζουν, ψηφίζουν, καταθέτουν τροπολογίες, αλλά τον ρόλο τον ενεργό, αν θέλετε, τον έχει στα χέρια του η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία. Και θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Όλα τα προβλήματα και οι δυσκολίες που υπάρχουν για την προστασία του καταναλωτή από αθέμητες εμπορικές πρακτικές περιέχουν και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη η οδηγία. Και γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και από νομικής πλευράς και από πρακτικής εφαρμογής του. Και πιστεύω ότι μία ενημερωτική εκστρατεία για τους καταναλωτές είναι πάρα πολύ, κάτι πολύ σημαντικό, διότι και στη χώρα μας υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, εμπορικές, ε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεν ξέρουν ότι μπορούν να στραφούν ε, σε μία αρχή για να ζητήσουν να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, και κυρίως όταν πρόκειται για ε, μερφοριακό εμπόριο, δεν ξέρουν πού να ζητήσουν βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την έννοια του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Προστασίας των Καταναλωτών για να διευκολυνθεί η προστασία των καταναλωτών. Αυτή, λοιπόν, αυτό το δίκτυο προστασίας των καταναλωτών πιστεύω ότι κάνει ποιοτική δουλειά και έχουμε ενωμερωθεί και για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε τώρα να μας μιλήσετε εσείς για την ε, θέση σε ισχύ της κοινοτικής οδηγίας του Αυτό το οποίο εμένα με εξέπλησε από τα σχόλια είναι το ότι τα διάφορα θέματα που αφορούν ε, τις διάφορες διασυνορικές πρακτικές δεν ε, αφορούν απευθείας στην εφαρμογή του νόμου. Πολλές φορές όταν δημιουργείται πρόβλημα μεταξύ Φερρυπίν, ε, Βελγίου και κάποιες άλλες χώρες, όλοι προσπαθούν να δούνε ποιος είναι ο νόμος που θα ισχύσει, Ποια είναι το δικαστήριο που θα δώσει την εγκατάλληλη εντολή. Χρησιμοποιούνται πολύ πολύπλοκα ε, νομικά επιχειρήματα για να δούμε αν είναι το βελγικό δίκαιο πρέπει να κάποιο άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προσκόμματα για να προχωρήσει κάποιο θέμα κανείς προστασίας από αθέμητες εμπορικές πρακτικές διασυνοριακώς. Και πολλές φορές οι άνθρωποι τα Τώρα εμείς σε μία περίπτωση ε, διαμάχης μεταξύ βελγικού και αγγλικού δικαίου πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά την συνεργασία ε, και που θα μπορούσε να υπάρχει οι βελγικές αρχές θα μπορούσαν να ασχοληθούν τις όλες επόθεσεις πιο εύκολα. Τώρα, ποιο είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο ε, πρέπει να ενεργήσει όταν οι δικοί του καταναλωτές στίγονται από μια πρακτική. Η λογική της ε, οδηγίας της δικαστικής εντολής ή διαταγής είναι κάτι το οποίο αφορά την δυνατότητα που δίνεται σε κάποιον από την δική του χώρα που έχει γίνει να προσφύγει δικά του δικαστήρια. Αλλά σε πολύ βασικό επίπεδο υπάρχουν ε, προβλήματα τα οποία ξεπερνούν κάποιον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να ζητήσει προστασία. Use, um, and legal Και βεβαίως Βεβαίω εδώ επισέρχονται και διάφορα οικονομικά θέματα και καλύτερα να είναι κανείς πολύ σωστά ενημερωμένος Κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι η εκπαίδευση των ε, εμπόρων. Πολλές φορές ο καταναλωτής ρωτά κάποιον υπάλληλο σε ένα έμπορο για τα ποια είναι τα δικαιώματά του, ο οποίος είναι ανενημέρωτος, τον οδηγεί σε... δεν τον ενημερώνει και τον οδηγεί σε παραπληροφόρηση καμιά φορά και μετά γίνονται τα πράγματα πιο πολύπλοκα και πολλές φορές από την παρανόηση μπορεί να δημιουργηθούν και περαιτέρω προβλήματα. Σωστά λέτε εσείς, δηλαδή, πρακτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει να υπάρχει στην πράξη δικαιοσύνη για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουν τον τέλειο τρόπο την ενημέρωση στους καταναλωτές για να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που μπορούν να εφαρμοστούν σε ιδιωτικές συναλλαγές, πώς θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν στα πλαίσια κέντρων ενημέρωσης προστασίας καταναλωτών, δικτύου προστασίας καταναλωτών. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και θα πρέπει να δούμε πώς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πιστούν να βοηθήσουν την επίλυση προβλημάτων που ξεκινάτων από τη δική τους χώρα. Thank you very much. We have Σας ευχαριστώ. Ε, And then, uh... Ευχαριστώ, δεν θα τα κάνεις το λόγο, στην οποία περίπτωση και θα ήθελα να καλύψουμε ίσως και άλλα, άλλες πτυχές της ε, προστασίας του καταναλωτή και να ακούσουμε και τη γνώμη σας για τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για αυτή τη σημαντική συζήτηση για τις συνθήκες της Λισαβόνας, θα δώσει όχι μόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερη εξουσία προκειμένου να συμμετάσχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Yes, one two. Who? Who? Baroness. Uh, Baroness. Um, It, I just thought it might be, um... Η Βαρόνη mm. Χάουαρτ από το Ενωμένο Βασίλειο. Um, I haven't asked a question because... Βαρόνη Χάουαρτ από το Ενωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται αυτή η διάδραση. Η διάδραση ό,τι αφορά το House of Lords. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία αποτελείται από αρκετές υποεπιτροπές, 80 είναι τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στην εξέταση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η δική μου επιτροπή είναι μία επιτροπή μόνο από αυτές που εξετάζουν τις διάφορες πτυχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να τονίσω, να παρέμβουμε σε αρχικό στάδιο και να υπάρχει αυτός ο έλεγχος όταν η οδηγία είναι σε αρκετά πρώτη αρχικό στάδιο. Και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπλοκές, ζητούμε μία έρευνα, το οποίο και σκοπεύουμε να κάνουμε με την προκειμένη οδηγία. Θα ήθελα να καλέσω και του συναδέλφου από τα άλλα κοινοβούλια να το εξετάσουν αυτό με πιο πολλή λεπτομέρεια, γιατί νομίζω ότι όσο πιο πολλέ λεπτομέρειε έχουμε για τον αντίκτυπο, γιατί αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο, ο αντίκτυπο για τους καταναλωτέ, ο αντίκτυπο της εναρμόνισης και κάποιε από τις ε, επιπλοκές του συμβατικού δικαίου. Αν είχαμε λοιπόν κάποια στοιχεία παραπάνω από άλλα κράτη, νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε για να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά να καταλήξει στην κατάρτιση μια σωστή οδηγία. που θα οθήσει και τις επιχειρήσεις αλλά και την πρόσταση των καταναλωτών. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, άλλες προτάσεις οι εμπειρίες που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Then my culture, we must, we must uh, exchange our opinion because we are in situation that we... Ναι, η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε χρόνο, αλλά μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ και την ε, συνάντησή μας μία ώρα νωρίτερα. Συμφωνείτε? Yes. Mm -hmm. Να περάσουμε λοιπόν στα καταληπτικά σχόλια. Και μετά, πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά διάλειμμα.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 Είναι μια πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική πραγματική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 aby se, aby se, aby to trošku jako tohle, já pak přečtu závěr, ještě budu jako už tohle, jo? Takže, And then you can invite at five o'clock. Yeah, yeah, I know. I know. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for your. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα συνεχίσουμε. The last uh, part of our session. Για το τελευταίο τμήμα της uh, συνάντησής μας. Θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω την, από την κυρία Παρκοντόβα να κάνει τα καταληκτικά της σχόλια. Κυρίε και κύριοι, και πάλι καλησπέρα σας. Μου ζητήθηκε να προσπαθήσω να συνοψίσω τη συζήτηση που δεν είχαμε. Ακούσαμε στο τελευταίο μέρος την ε, ομιλία του Άγγλου προσκεκλημένου μας, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν θα κάνω κανένα σχόλια, αλλά πρέπει να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο, η, ο έλεγχος και για την μεταφορά της οδηγίας, έτσι όπως ε, την ε, κάνει η Βουλή των Λόρδων, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρον. Πρέπει να πω ότι εμείς στη χώρα μας έχουμε διαφορετικό τρόπο και διαπιστώνουμε ότι σε κάθε εθνικό επίπεδο είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ε, το όλο θέμα της προστασίας των καταναλωτών ε, ε, ισχύει. Θα ήταν πολύ εύκολο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους να κάνουμε λοιπόν μία συγκριτική ανάλυση, να δούμε επίσης τι προβλέπει ο κάθε αστικός κώδικας και ακόμη να συμπεριλάβουμε και στον αστικό κώδικα, ε, ε, κώδικα κάθε κράτους ε, τα δικαιώματα, τα βασικά των καταναλωτών. Πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια της παρούσης προεδρίας μας αυτό το θέμα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο. Χρήσιμο το ότι ασχολήθηκαν οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να ασχοληθούν και όλοι οι συνάδελφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Βεβαίως, Πιστεύω ότι μετά από την θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας θα μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις συναντήσεις μας και την um, anybody... Να σας ζητήσω τα σχόλιά σας, αν δεν συμφωνείτε. Έχετε πάντα δυνατότητα να μας ε, βελτιώσετε. Η κατάτμιση της ε, νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών αποτελεί μια ανησυχία και αυτό τονίστηκε στις, ε, στις πιο πολλές ε, παρεμβάσεις ό,τι αφορά και την τρέχουσα οικονομική κρίση. Μόνο μια σωστά και έμπριθμα λειτουργούσα ενιαία αγορά μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση ε, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται. Μία γενική ομοφωνία, συνένεση για την ε, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων ακούστηκε από πολλές ε, παρεμβάσεις και η ευρωπαϊκή εναρμόνιση αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ένα σημαντικό βήμα σημειώθηκε σήμερα, από ό,τι φαίνεται, οι πιο πολλοί συμμετέχοντες συμφωνούν για τους στόχους της πρότασης αυτής και για την ανάγκη ύπαρξης εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε όλες τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης τονίστηκε. Κάτι άλλο, ότι η σωστή αξιολόγηση των, της πλήρους εναρμόνισης θα πρέπει να γίνει προτού προχωρήσουμε περαιτέρω. Εν γέννη, οι συμμετέχοντες ζήτησαν να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους όρους και το πεδίο εφαρμογής. Ζήτησαν καλύτερη κατανόηση μεταξύ της σχέσης που έχει και της σύνδεσης αυτής της νομοθεσίας με τις άλλες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωση. σε ό,τι αφορά τους συμβατικούς όρους και τους αθέμετους όρους. Η Επιτροπή ΕΜΚΟ συμφωνεί με τις ανησυχίες αυτές, τις οποίες και θα λάβει δεόντως υπόψη όταν θα εξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις εργασίες, ε, τις μελλοντικές ε, της ε, Επιτροπής ΕΜΚΟ ένα σχέδιο, ένα έγγραφο εργασία θα καταρτιστεί μέχρι τα τέλη τη εβδομάδα και θα διανεμηθεί και ασφαλώ στη Εθνικά Κοινοβούλια για σχόλια. Έχετε κάποιο σχόλιο? Do agree with this uh, Συμφωνείτε με αυτές τα σχόλια, τα καταληκτικά, τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους ε, εισηγητές ε, των εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας. Θα υπάρξουν κατά πάσα πιθανότητα πάρα πολλές τροπολογίες για την οδηγία αυτή. Κατά την επόμενη εκλογική περίοδο. Είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω ότι την επόμενη φορά θα δούμε. Ότι θα σας ξαναδούμε λοιπόν όλους και θα ήθελα να σας καλέσω στο κοκτέιλ μας. Ζητήσαμε Προετοιμαστεί το κοκτέιλ αυτό στις 5 και όχι στις 6. Μπροστά από την αίθουσα. Επειδή δεν υπάρχουν ερωτήσεις ε, για τη μεταφορά της οδηγίας. Μόνο οι κυρίες από την Τσεχική Δημοκρατία. Yeah. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας.